morning. Good morning. Καλημέρα σας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. It is also today the morning session and the afternoon session. So Έχουμε πρωινή και απογευματινή συνεδρία με φορτωμένη μερική διάταξη. Περνάμε στο σημείο υπαριθμών 21 που είναι το πρώτο σημείο το οποίο προβλέπεται για σήμερα το πρωί σε σχέση με τη δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Please, let me first go through the announcements. Να κάνω πρώτα τις ε, ανακοινώσεις. το σχέδιο χρονοδιαγράμματος των συνεδριάσεων της ΛΥΜΠΕ για το 2013. Έχει εγκριθεί από τους συντονιστές το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεών μας για το 2013. Ελήψη ενστάσεων θα θεωρηθεί ότι έχει εγκριθεί. Μετά έχουμε το θέμα του διορισμού εισηγητών. Η κυρία Ρενάτε Ζόμερ από το ΕΛΚ είναι εισηγήτρια για την συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας για την επανεισδοχή ατόμων χωρίς έγγραφα διαμονής. Και συντάκτης γνωμοδότησης ο κύριος Γιάνς Μπρόντε από την ομάδα ALDE, συντάκτης γνωμοδότησης για την έκθεση ηλεκτρονικές υπηρεσίες ταυτοποίησης και δημιουργίας εμπιστοσύνης για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο κύριος Μπουσούτιλ από το ΕΛΚ θα είναι και ο συντάκτης γνωμοδότησης για την ε, εφαρμογή της ε, ρήτρα άμυνας και αλληλεγγύης. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις που ήθελα να κάνω και χρειάζομαι την ε, έγκριση της Επιτροπής. Τούτου λεχθέντος περνάμε στο σημείο υπαριθμών 21 το Δεκέμβριο του 2011 το Κοινοβούλιο <clears throat> ενέκρινε την ε, θέση πρώτης ανάγνωσης για την αναδιατύπωση οδηγία σε σχέση με τη δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα. Έχουν λάβει χώρα διάφοροι τριγωνικοί διάλογοι κατά τη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας. Μάιο-Ιούνιο του 2012 έχουν λάβει αυτές οι συναντήσεις. Παρά τις προσπάθειες όμως του εισηγητού μας εδώ, του κύριου Κάσμαν, μαζί με την Δανική Προεδρία δεν έχει επιτευχθεί καμία συμφωνία για το θέμα αυτό. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον εισηγητή μας ο οποίος θα μας παρουσιάσει την κατάσταση πραγμάτων μετά τους τριγωνικούς αυτούς διαλόγους. Κύριε Κάσμαν, σας ευχαριστώ. Λέω Κάσμαν. Καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους. Δεν πρόκειται να χρονοτριβήσω ιδιαίτερα γιατί νομίζω ότι <clears throat> οι περισσότεροι σκιώδεις εισηγητές γνωρίζουν την κατάσταση όπως και αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν από κοντά το θέμα. Όπως σωστά είπατε, η Δανική Προεδρία είχε μία εντολή από το Συμβούλιο και επί τη βάση αυτής διαπραγματευτήκαμε για ένα κατάλογο 10 σημείων. Αλλά πρέπει να πω ότι και εγώ και οι υπόλοιποι εισηγητές χάρηκαν ιδιαίτερα και διαφωτίστηκαν από την προσέγγιση της Δανικής Προεδρίας. Μετά περάσαμε σε ομάδε εργασία σύνταξη, όπου και πάλι φάνηκε να υπάρχει κάποια πρόοδο. Αλλά εν τέλει και τελικά η Δανική Προεδρία επιζήτησε μια άλλη εντολή από το Συμβούλιο, μια διαφορετική εντολή που το Συμβούλιο τη απέρριψε, δεν τη έδωσε τέτοια εντολή. Προχωρήσαμε λοιπόν <clears throat> σε μια σύγκληση για ορισμένα θέματα που μπορώ να αναφέρω σε λίγο. Ο Μαρκ Μέιζ από την Κομισιόν ελπίζω να μην το πάρει προσωπικά αυτό που θα πω. Αλλά εγώ θα πρέπει να πω ότι αν δεν ήταν η Κομισιόν θα μπορούσαμε να είχαμε καταλήξει σε μια συμφωνία με την Δανική Προεδρία. Το κατά πόσο τώρα το Συμβούλιο θα είχε δεχτεί ή όχι αυτή η συμφωνία είναι τελείως διαφορετικό θέμα. Πρέπει να πω επίσης ότι στα πλαίσια της σύνταξης προσπαθώντας να επιλύσουμε ορισμένα προβλήματα ο ορισμός του τι είναι έγγραφο στην προσπάθεια να έχουμε μια πιο περισταλτική ε, η Κομισιόν προσπαθούσε να έχει μια πιο περισταλτική ε, θέση στο τι αποτελεί έγγραφο για να μειώσει και την πρόσβαση. Επομένως, ακόμα και η δυνατότητα διαπραγμάτευση με την Προεδρία ήταν περιορισμένη μετά από όλα αυτά. Πρέπει να σα πω επίση, και αυτό πάλι είναι κάτι το οποίο έχω πει δημόσια στον παρελθόν, σε καμία χρονική στιγμή, μετά από τι αιτήσει μου εξ του Κοινοβουλίου και μετά από τι αιτήσει τη Δανική Προεδρία, όταν είπαμε στην Κομισιόν <clears throat> ότι αν έχουν προβλήματα θα πρέπει να προτείνουν συντακτικές λύσεις σε καμία χρονική στιγμή η Κομισιόν δεν μας έφερε προτάσεις σύνταξης στην ομάδα εργασία σύνταξης ή τέσσερα περαιτέρω συναντήσεις. Όλα αυτά δεν με εκπλήσουν γιατί ξέρω ότι η Κομισιόν έχει ακολουθήσει μια πολύ διαφορετική και περιοριστική άποψη σε σχέση με την πρόσβαση στα έγγραφα από ό,τι που ακολουθώ εγώ και οι περισσότεροι συνάδελφοί μου. Τα σημεία στα οποία υπήρξε σύγκληση απόψεων και εδώ αναφέρομαι στα σημειώματά μου ορισμός του στόχου της, ε, του κανονισμού, η αναφορά σε καλές διοικητικές πρακτικές, η τωρινή κατάσταση στα κράτη-μέλη που δεν θεωρούνται τρίτες χώρες. Καλό θα ήταν να μην με διακόπτουν ορισμένοι οι οποίοι κάνουν πηγαδάκια όταν προσπαθώ να παρουσιάσω αυτό το θέμα. Εγώ χαίρομαι να ακούω τους άλλους, αλλά ναι, παρακαλώ. Ο Μάικλ Κάσμαν ζητάει να έχει την προσοχή σου. Όχι για σένα, Μόνικα. Όταν κάποιος έχει το λόγο όμως, ιδίως όταν υπάρχουν πολίτες και ΜΚΟ στην αίθουσα που παρακολουθούν τις εργασίες μας, δίνει το λανθασμένο μήνυμα όταν οι άλλοι δεν τον ακούν. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να με ακούν οι πολίτες. Διευκρίνηση λοιπόν για κάποια κράτη-μέλη που δεν θέλουν τρίτες χώρες όταν λειτουργούν σαν μέλη του Συμβουλίου ή όταν εξετάζονται κατ' εξουσιοδότηση πράξης. Επέκταση της σφαίρας εφαρμογής σε όλα τα δεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και αποκεντρωμένους φορείς και γραφεία. Η νομοθετική διαφάνεια, η εισαγωγή γραφείων πληροφόρησης και καταληκτικές προθεσμίες για την διεκπαιρέωση των αιτήσεων. Κάτι λοιπόν το οποίο δεν αποτέλεσε αντικείμενο συμφωνίες <clears throat> ήταν το θέμα της ανησυχηρίας που μπορεί να προταθεί από ένα κράτος μέλος και εκεί η Ιδανική Προεδρία είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία δυνατότητα βέτο από ένα κράτος μέλος. Αλλά είπε το εξή, ότι για να εξηγήσουμε γιατί υπάρχει μια εξαίρεση, ένα κράτο μέλο μπορεί να αναφερθεί σε οποιασδήποτε σχετικέ ρήτρε ή κανόνε στην εθνική του νομοθεσία. Όπω λέει ο κανονισμό, ο κανονισμό για την μη πρόσβαση στα έγγραφα μπορεί να βασίζεται μονάχα σε αυτά τα οποία λέει το άρθρο 4 και το άρθρο 9. Το να υπάρχει μια τέτοια ρήτρα θα έδινε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη <clears throat> να ξεπεράσουν ουσιαστικά τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού ιδίως για την θέση ενός κράτους μέλους στο Συμβούλιο. Επίσης τα θέματα για νομική ε, αρρωγή και πυρογνωμοσύνη δεν προχωρήσαμε για αυτά τα οποία θεωρούνται συνολικές εξαιρέσεις και όλα αυτά δεν έχουμε καταλήξει λύση. Εγώ συζήτησα με την Κυπριακή Προεδρία, με εντυπωσίασε η ενεργητικότητα και ο ενθουσιασμό του στο θέμα αυτό. Είχαμε μια άτυπη συνεδρίαση όπου εκφράσαμε τη θέλησή μας να προχωρήσουμε στα θέματα αυτά. Αναμένω ακόμα να δω αν υπάρχει κάποια επίσημη εντολή από το Συμβούλιο προς την Κυπριακή ε, Προεδρία, αν είναι η ίδια όπως το σχέδιο 10 σημείων που είχαμε στην ε, Δανική Προεδρία. Αν είναι αυτό το ίδιο θα ξαναγυρίσουμε στο σημείο κίνησης, αλλά πρέπει να υπάρξει κάποια κίνηση για τα θέματα αυτά. Εγώ βλέπω η Κομισιόν να τροχοποδεί τροχοπεδί το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και να μην τους επιτρέπει να καταλήξουν σε κάποια λύση αυτή τη στιγμή. Διατηρώ τις ελπίδες μου παρόλα αυτά ότι μπορούμε να επιτύχουμε κάποια πρόοδο <clears throat> κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας διότι έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία και έχουν δείξει μεγάλη προσήλωση στην επίλυση αυτών των θεμάτων. Κλείνω εδώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τη σύνοψη και για όλη την εργασία που έχετε κάνει για το θέμα αυτό. σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Μετά από τον κύριο Κάσμαν, υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να λάβει το λόγο, κάποιος θέλει να σχολιάσει, κύριε Κάσμαν. Ίσως πρέπει να περάσετε το λόγο στην Προεδρία, οι οποίοι είναι παρόντες εδώ το πρωί και ίσως και η Επιτροπή να έχει κάποια απάντηση ε, στην πρόκληση θα έλεγα την οποία τους απίφθηνα σήμερα εκπρόσωπος του Συμβουλίου παρακαλώ μπορείτε να συστηθείτε πρώτα Παρακολουθώ το θέμα αυτό εδώ και αρκετό καιρό. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να είμαστε εδώ σήμερα. Ακούσαμε προσεκτικά αυτά που είπε ο κύριος Κάσμαν. Να τονίσω το εξής. Το θέμα είναι σημαντικό. Είναι περίπλοκο και θα θέλαμε εμείς να συνεχίσουμε να έχουμε στενές επαφές και με τον εισηγητή και με το κοινοβούλιο. Ξεκινήσαμε το καλοκαίρι τις άτυπες επαφές με τον κύριο Κάσμαν και θα συνεχίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση τις επόμενες εβδομάδες. Έχει γίνει σημαντική δουλειά κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Δανίας και υπήρξε πρόοδος σε σημαντικά θέματα που εξήγησε άλλωστε ο κύριος Κάσμαν. Υπάρχουν διαφορές σε ορισμένα σημεία βέβαια, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να γεφυρώσουμε τις διαφορές με ρεαλιστικές λύσεις. Εμείς θα βασιστούμε στην πρόοδο η οποία έχει σημειωθεί και καλό θα είναι να σημειώσει κανείς την εξαιρετική δουλειά που έκαναν οι Δανείοι. Θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις και με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη στα πλαίσια της ομάδας εργασίας για την πληροφόρηση. Εποφελούμενος από αυτά που είπε ο κ. Κάσμαν για την Επιτροπή και τα λοιπά, θα πρέπει να τονίσω, και αυτή είναι η αίσθησή μου από τις αρχικές επαφές, η αίσθησή μου είναι ότι ο φάκελος αυτός απαιτεί περισσότερο χρόνο Πρέπει να οριμάσει κάπως η κατάσταση ώσπου να βρούμε αυτές τις ε, λύσεις που αναζητούμε. Εμείς σαν Κυπριακή Προεδρία εκτιμούμε λοιπόν τις συζητήσεις που ξεκίνησαν με τον κύριο Κάσμαν, θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις αυτές και σημειώνω εδώ και την ευελιξία και την καλή βούληση, καλή θέληση που εξέφρασε ο κύριος Κάσμαν σήμερα και θα τον διαβεβαιώσω ότι θα την εκμεταλλευτούμε κατάλληλα. Ένα τελευταίο σημείο. Θα χρησιμοποιήσω την παραδοσιακή ελληνική σοφία. Θα ακολουθήσουμε λοιπόν το σπέβδε βραβέως. Ευχαριστούμε την Προεδρία. Εκπρόσωπος της Επιτροπής τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τεγλή αναφέρομαι, ναι, ονομάζομαι από την ε, Γενική Γραμματεία της Επιτροπής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, και εγώ τη Δανική Προεδρία για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει για να προχωρήσει αυτό το δύσκολο θέμα. Θα ήθελα επίσης να συμφωνήσω με τις ευχές που εκφράστηκαν και ελπίζω και εγώ η Κυπριακή Προεδρία να συνεχίσει με, αυτό, με αυτή την ε, καλή θέληση που έχει ξεκινήσει. Ακούσαμε τις ε, παρατηρήσεις του κυρίου Κάσμαν. Βεβαίω εδώ τώρα δεν έχουμε έρθει ούτε για να ε, έρθουμε σε αντιπαράθεση, ούτε για να μιλήσουμε επί της ουσίας αυτής της πρωτοβουλίας. Θα ήθελα βεβαίως να επιβεβαιώσω ότι εμείς ως Επιτροπή επιθυμούμε να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή συμφωνία ε, για ένα θέμα που αφορά την προστασία των ίδιων των πολιτών. Αποδίδουμε μεγάλη σημασία λοιπόν στην ικανοποίηση των ε, αναγκών των πολιτών. Ε, Βεβαίω είναι περίπλοκο το θέμα λόγω των διαφόρων συμφερόντων που υπάρχουν και γνωρίζετε και γνωρίζουμε ότι τα, τα ευρωπαϊκά όργανα ε, έρχονται αντιμέτωπα κάθε μέρα με το περιπλοκότητα του ζητήματος, ε, με διαφορετικές μορφές ε, κειμένων και γράφων και το καθεξής. Ξέρουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία. Η Επιτροπή θα κάνει ό,τι μπορεί για να διευκολύνει την ανάδειξη της καλύτερης δυνατής συμφωνίας. και είμαστε μάρτυρες και είστε μάρτυρες ε, της σκληρής προσπάθειας που έχει καταβληθεί από τις υπηρεσίες μας για να καταλήξουμε στην ε, καλύτερη δυνατή διατύπωση στο κείμενο. Μπορώ λοιπόν ε, επισήμως να πω ότι η πρόταση που έγινε από την Επιτροπή στην αρχή ούτε ήταν, ούτε είναι, ούτε θα είναι βήμα προς τα πίσω ε, σε ζητήματα διαφάνειας. Ε, το έχουμε εξηγήσει, είμαστε διεθμένοι να το κάνουμε και στο μέλλον. Να εξηγήσουμε λοιπόν ε, τα κίνητρα της πρότασής μας που λαμβάνει υπόψη την ομολογία, την πρακτική ε, λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των ε, πολιτών και μπορούμε να βασιστούμε σε συγκεκριμένες ε, υποθέσεις. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν θα αποτελέσει βήμα προς τα πίσω. Ε, επαναλαμβάνω ότι κάθε έγγραφο που σε αυτό το αρχικό στάδιο μπορούν να δημοσιευθούν βάσει του 1049 θα γίνεται αυτό με τον ίδιο τρόπο όπως την πρότασή μας. Ευχαριστούμε την Επιτροπή. Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις. Ή να δώσουμε το λόγο και πάλι στον κύριο Κάσμαν. Παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα, ένα ερώτημα προς την Προεδρία. Τι μας λένε ουσιαστικά, ότι δεν προβλέπεται τριμερής διάλογος. Θα υπάρξει κάποιο χρονοδιάγραμμα γιατί δυστυχώς έχετε ακόμα 3,5 μήνες, μην σας πω και λιγότερο, στην εξαιρετική σας Προεδρία. Άκουσα και τον εκπρόσωπο της ε, Επιτροπής. Νομίζω ότι με πολύ όμορφο τρόπο μας είπε γιατί δεν μπορούμε να καταλήξουμε στη συμφωνία. Είπε ότι τώρα, σήμερα το πρωί, η πρωινή συνεδρίαση δεν είναι μια καλή ευκαιρία για να έρθουμε στην παράθεση. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς με το να λέει κανένα ότι όσοι γνωρίζουν το θέμα καλά είναι μάρτυρες ε, ε της προσπάθειας Επιτροπής να καταλήξει στην καλύτερη δυνατή διατύπωση. Δεν έχει ακούσει η Επιτροπή τη Μη κυβερνητική οργανώσεω από την αρχική πρόταση που την ε, καταδίκασαν. Ε, ο Ευρωπαίος Επόπτη Προσωπικών Δεδομένων, ο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τόσοι οργανισμοί που μας είπαν ουσιαστικά ότι η ερμηνεία που δίνεται δεν υπηρετεί τα συμφέροντα των ε, ε, πολιτών. Επίσης, ε, χρησιμοποίησα τον όρο προστασία των πολιτών. Συμφωνούμε βεβαίως με αυτό. Αλλά αυτό αναφέρεται στο άρθρο 4 και 9, στις εξαιρέσεις. Αν θέλετε συνεκτική προστασία της εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας, μαζί με άλλα ζητήματα βεβαίως που απασχολούν τους πολίτες μας, τότε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, ε, η Συνομική Επιτροπή, θα αποδεχθούν τη θέση του Κοινοβουλίου ότι χρειαζόμαστε κοινού κανόνε ταξινόμησης και στα τρία όργανα, ούτω ώστε κάθε όργανο να ε, αποδέχεται και να αναγνωρίζει την ταξινόμηση ε, που δίνεται από το άλλο. Αν δεν συμβαίνει αυτό, τότε υπονομεύεται η προστασία των ε, συμφερόντων. Ανέφερε ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή ότι είναι καλύτερη δυνατή συμφωνία για ποιον είναι αυτή η καλύτερη δυνατή συμφωνία. Ε, βάσει της δικής μας μελέτης και ε, βάσει της ε, αγγλικής γλώσσας και της γνώσης μου αυτής, οι ορισμοί υπονομεύουν το τρέχον εφιστάμενο επίπεδο πρόσβασης και διαφάνειας. Η Επιτροπή είπε ότι οι παρατηρήσεις μου αναφέρθηκε σε παρατηρήσεις που έκανα σήμερα το πρωί. Είναι πράγματι, είναι παρατηρήσεις και όπως όλες οι παρατηρήσεις μπορούν να είναι μονομερείς. Επομένως, ε, δεσμεύομαι ενώπιον τη Επιτροπής και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα δημοσιεύσω ε, τις ε, διάφορες προτάσεις της Προεδρίας και, που, και τις προτάσεις που δεν ήρθαν από την Επιτροπή και οι συνάδελφοι που λένε ότι θα πούνε ότι οι παρατηρήσεις μου βασίζονται σε ε, αποδεικτικά στοιχεία, αν θέλετε. Και αν ε, κάποιος ε, μπορεί να αποδείξει το αντίθετο, θα τις αποσύρω. Είναι ένα πολύ καλό, ένας πολύ καλός Το πολύ καλό στοιχείο για τους πολίτες μας και για το Κοινοβούλιο είναι ότι εγώ και άλλοι εδώ στο Κοινοβούλιο δεν πρόκειται να υπονομεύσουν την υφιστάμενη πρόσβαση στα έγγραφα. Δεν θα μειώσουμε τα δικαιώματα των πολιτών μας, γιατί μεσούς της κρίσης ε, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο πρέπει να εξηγήσουμε περισσότερο τι κάνουμε εδώ ε, και όχι λιγότερο. Αλλιώς ε, οι πολίτες θα μας γυρίσουν την πλάτη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κάσμαν. <clears throat> Ξέρουμε ότι ο κύριος Κύρκοφ θέλει να κάνει ένα σύντομο σχόλιο τώρα. Του δίνω λοιπόν το λόγο και μπορεί να χρειαστεί να επανέλθετε κύριε Κάσμα, κύριε Κύρχοφ. Δεν νομίζω θα χρειαστεί να απαντήσει σε μένα κύριο κύριος Κύρκοφ και ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα να έρθω. Παρακολούθησα μονάχα τα τελευταία λεπτά μιας παρουσίασης πενταετούς οικονομικού σχεδίου σοβιετικού χαρακτήρα από την Κομισιόν. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά, αλλά δεν αντιμετώπισε τα προβλήματα που ανέφερε ο κύριο Κάσμαν για να είμαστε σαφείς, θέλω να, τονίσω ότι υποστηρίζω ιδιαίτερα τη θέση του κυρίου Κάσμαν και νιώθω κάποια απογοήτευση από τις ε, κάπως υποτιθέμενες παρατηρήσεις ορισμένων θεσμικών οργάνων σε σχέση με το θέμα αυτό. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και υπάρχουν πολλές προσδοκίες από τους πολίτες της Ευρώπης, κύριε Πρόεδρε, και εγώ συνεχίζω να υποστηρίζω διαρρήνη τον κύριο Κάσμαν και η δική μου πολιτική ομάδα και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μία πρόοδο. Όλοι υποστηρίζουμε τον Μάικελ Κάσμαν ως εισηγητή για το θέμα αυτό, το οποίο έχει χρονίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και Κάσμαν. Δεν θέλω να θέσω σε δύσκολη θέση τους Κύπριους ε, συναδέλφους μου, αλλά θα ήθελα απλώς να ξέρω αν προβλέπουν μέσα στο χρονοδιάγραμμα αυτό κάποια δυνατότητα λύσης για αυτά τα προβλήματα. Η Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. 3,5 μήνες είναι επαρκής χρόνος κατά τη δική μου άποψη για τα επόμενα βήματα όμως που θα πρέπει να ληφθούν. Εμείς ελέγχουμε τις δυνατότητες που έχουμε. Είναι προφανές ότι προσπαθούμε να βρούμε κάποιο χώρο, κάποιο περιθώριο ενεργειών και βάσει των στοιχείων που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε χωρίς να αποκλείσουμε φυσικά τη δυνατότητα να λάβει χώρα ένας ε, άτυπος ε, τρίλογος εν καιρό ή μια οποιαδήποτε άλλη μορφή συνεδρίαση. Αλλά προς το παρόν πρέπει να σας αναφέρω ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα περιθώριο ελιγμών και θα παραμείνουμε σε στενή επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, όχι, λέει ο κ. Κάσμαν. Εντάξει, λοιπόν, σας ευχαριστούμε για την πληροφόρηση και τη σύνοψη που μας έχετε παρουσιάσει και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης για την επόμενη μισή ώρα. Το σημείο 7 για το πάγωμα και την κατάσχεση προϊόντων εγκλημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Μόνικα Μακοβέη είναι η για το θέμα αυτό. Γνωρίζετε όλοι ότι το θέμα που μας απασχολεί εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι για την ε, αντιμετώπιση των προσόδων από το έγκλημα. Ο κόσμος μας, ο παγκοσμιοποιημένος, περιστρέφεται και περισσότερο από το χρήμα, αλλά και το παγκοσμιοποιημένο χρήμα και έχουμε ενώπιον μας μια πρόταση οδηγίας για την ε, κατάψυξη και την κατάσχεση των εσόδων από εγκληματικές ενέργειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι μια καλόδεκτη πρόταση στην, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί ανταποκρίνεται σε αυτά τα οποία ανέφερε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ένα ψήφισμα το οποίο είναι τον Οκτώβριο του 2011 ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οργανωμένο έγκλημα. Η πρόταση αυτή λοιπόν <clears throat> θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης, θα δώσει ένα νομικό πλαίσιο με νέους κανόνες για ε, επέκταση των, δυνατό, δυνατοτήτων κατάσχεσης, κατάσχεσης που δεν έλκεται μόνο από καταδίκη, καταδίκη υπέρ τρίτου και κατάψυξη στοιχείων ενεργητικού που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν ή να παροχετευτούν σε άλλες κατευθύνσεις. Ένα σύνολο λοιπόν από <clears throat> πρόνοιες που αφορούν την ανάγκη να διαφυλάξουμε αυτά τα έσοδα από εγκληματικές ενέργειες. Τα κάτι μέλη ως εκ τούτου θα είναι υποχρεωμένα να διαχειρίζονται κατάλληλα τα κατεψυγμένα αυτά έσοδα ώστε να μην χάνουν την οικονομική τους αξία πριν από την οριστική τους κατάσχεση. Έχουν λοιπόν να κάνουν τη διαχείριση αυτών των στοιχείων ενεργητικού. Η κυρία Μόνικα Μακοβέη θα μας παρουσιάσει λοιπόν το θέμα αυτό και θα ακολουθήσει μετά ο καθορισμός μιας καταληκτικής προθεσμίας για τις τροπολογίες. Κύριε Μακοβέη, σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για μια ακόμη φορά ζητώ συγγνώμη, δεν είναι εδώ ο κύριος Κάσπμαν, βλέπω, θα του το μεταφέρω. Ευχαριστώ για την εισαγωγή που κάνατε και εγώ πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να παρακολουθεί κανείς τα χρήματα που παράγονται από εγκληματικές δραστηριότητες και αυτό είναι πολλές φορές πιο σημαντικό από το να στείλει κάποιον κάποιοι σε φυλακή γιατί ε, τα οικονομικά μέσα είναι αυτά τα οποία άμα ελείψουν θα τους παρεμποδίσουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και θα τους εμποδίσουν να περάσουν σε άλλες παράνομες δραστηριότητες όπως η έκπληνση δρομικού χρήματος. Η πρόταση της Επιτροπής έγινε δεκτή τον μήνα Μάρτιο. Καθορίζει τους μίνιμουμ κανόνες για το πάγωμα και την κατάσχεση των προϊόντων εγκλήματος. Παρατεταμένη κατάσχεση, ε, κατάσχεση που δεν βασίζεται σε απόφαση δικαστηρίου και κατάσχεση ε, ιδιοκτησιών ε, τρίτων πλευρών. Θα ήθελα να πω ότι η υιοθέτηση όλων αυτών των κανόνων θα βελτιώσει τις νομικές συνθήκες στα κράτη-μέλη, θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη και θα ενισχύσει στον τομέα τον ποινικό και την σωστή συνεργασία. Στόχος μου είναι να ενισχύσουμε τις κατασχέσεις ε, ε, που δεν βασίζονται σε απόφαση δικαστηρίου, τις κατασχέσεις τρίτων πλευρών ή τις κατασχέσεις παρατεταμένης διάρκειας έτσι ώστε να αστερίσουμε τα μέσα και να μην μπορέσουν να προχωρήσουν σε περαιτέρω παράνομες δραστηριότητες όπως το μη νόμιμες. Uh, my proposal on the non-conviction based confiscation όπως η έκπληνση χρήματος and provide for confiscation of proceeds and instrumentalities of crime in civil proceedings for Εδώ θα ήθελα λοιπόν να ενημερώσω τους παρισταμένους και βλέποντας και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπάρχει μία απόφαση του δικαστηρίου αυτού, η απόφαση Μπάτλερ, εναντίον Ηνωμένου Βασιλείου. Η απόφαση αυτή λέγει ότι οι κατασχέσεις που δεν βασίζονται σε δικαστική καταδίκη στα πλαίσια του αστικού δικαίου ε, είναι κάτι το συμβατό με το ευρωπαϊκό δίκαιο εφόσον γίνεται με νόμιμο τρόπο και εφόσον υποστηρίζεται και έχει κανονική υπεράσπιση από δικηγόρο κατηγορούμενο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρεί ότι τέτοιου είδους αστικές διαδικασίες εντάσσονται στα δικαιώματα των κρατών μελών να επιβάλλουν συγκεκριμένες νομικές ρυθμίσεις και να ελέγξουν τη χρήση της ιδιοκτησίας ε, προς το γενικότερο όφελος. Αυτό παραπέμπει λίγο στο ερώτημα το οποίο έχει τεθεί από ορισμένου συναδέλφους γύρω από την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τώρα, το θέμα της κατάσχεσης μέσω αστικών διαδικασιών στην περίπτωση δραστηριοτήτων ποινικού τύπου είναι κάτι το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε ορισμένες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Ιταλία, Σλοβενία, Σλοβακία και στις Ηνωμένε Πολιτείε φυσικά από όπου και ξεκίνησε. Θα ήθελα εκ των προτέρων να πω ότι οι αλλαγές που θα κάνω στην έκθεσή μου είναι οι εξής, έτσι θα σας γλιτώσω τροπολογίες και χρόνο. Θα ήθελα να αποσύρω την τροπολογία 5 σχετικά με τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σε ποινικέ πράξεις οι οποίες μπορεί να τιμωρηθούν με μέγιστη διάρκεια φυλάκιση στο ένα έτος. Και θα κρατήσω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία περιορίζει την εμβέλεια και εφαρμογή της ρύθμισης στο οργανωμένο έγκλημα όπως περιγράφεται στην παράγραφο, στο άρθρο 83 παράγραφος 1. Αποσύρω τις τροπολογίες 12 και 14 σχετικά με τον αποκλεισμό της μεθόδου της ε, διευρυμένης κατάσχεσης εφόσον έχει αθωωθεί το συγκεκριμένο πρόσωπο. Στην περίπτωση που έχει υπάρξει αθώωση σε επίπεδο ποινικό δεν θα πρέπει να είναι δυνατόν να υπάρχει κατάσχεση μέσω μιας αστικής διαδικασίας για τη συγκεκριμένη ποινική ενέργεια. Οπότε σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζεται ο νόμος ως έχει. Το να αντιπροσωπεύεται κανείς από δικηγόρο είναι κάτι το οποίο είναι αντικείμενο εγγύησης από τις Ευρωπαϊκές Συμβάσεις και θα επανέλθει στο κείμενο μετά από συζητήσεις που είχαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταλήξουμε σε μια διατύπωση η οποία θα είναι πιο ξεκάθαρη και όποιος έχει τα χρήματα να πληρώσει δικηγόρο μπορεί να το κάνει και τα κρατη δεν θα είναι ε, υποχρεωμένα εξοφίκιο να παρέχουν ε, δικηγόρο νομική προστασία. Για το χρονοδιάγραμμα τώρα. Το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Η πρότασή μου λοιπόν είναι να γίνει η παρουσίαση της πρότασης σήμερα, όπως ακριβώς συμβαίνει 9 Οκτωβρίου προθεσμία κατάθεση τροπολογιών και πιθανή παρουσίαση των τροπολογιών στις διάφορες πολιτικές ομάδες ή τις συναντήσεις των σκιωδών. Η προσανατολιστική ψηφοφορία μπορεί να γίνει στη συνεδρίασή μας στις 27 Νοεμβρίου. Εν τω μεταξύ και για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες θα έχω ήδη συναντηθεί με τους σκιώδεις εισηγητές, προχθές μάλλον συναντήθηκα με τους σκιώδεις εισηγητές, χθες συγγνώμη, Είμαι βέβαιος ότι μετά τη συνάντηση αυτή, είμαι βεβαία ότι θα βοηθήσουν για να γίνει καλύτερη η έκθεση αυτή. Ευχαριστώ κυρία Μακοβέη. Πριν δώσουμε το λόγο στους βουλευτές, θα δώσουμε το λόγο ίσως στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριο Σπρίμπκε, και μετά εάν θέλει η Προεδρία. και μετά στα μέλη τα οποία έχουν πει ότι ενδιαφέρονται να πάρουν το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επιτροπή για την στήριξή της και ιδίως προς ε, την εισηγήτρια για την ε, πρόταση της Επιτροπής με το πάγωμα για τη δίμευση. Πράγματι, η απάντηση της Επιτροπής για το επίγον αίτημα για νομοθέτηση ε, πράξης ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση μας βρίσκει σύμφωνος. Πράγματι, είναι ε, έκτακτο το ζήτημα αυτό. Το σχέδιο έκθεσης ε, υπογραμμίζει την ανάγκη τη αύξηση τη αποδοτικότητα του νέου νομοθετικού πλαισίου και εμεί Είμαστε ανοιχτά διακείμενοι απέναντι στις ε, διάφορες τροπολογίες που έχουν ε, που έχουν κατατεθεί ε, και θα βοηθήσουν τη διαδικασία της κατάσχεσης των προσόδων του εγκλήματος κάποια σημεία για την ε, τροπολογία 4. Προτείνεται η εισαγωγή ε, συστήματος ε, δίμευσης που δεν βασίζεται στην καταδίκη, όπου η δίμευση μπορεί να γίνει και ελλείψη προσόδων από εγκληματικές πράξεις. <clears throat> Αυτό μπορεί να γίνει όταν η δίεξη δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ή να συνεχιστεί. Η τροπολογία 4 λοιπόν ε, ξεφεύγει από το ε, πεδίο της ε, πρότασής μας μετά στην 23. Όταν είναι χαμηλότερη της αξίας αγοράς, αυτό επηρεάζει τα δικαιώματα καλή πίστη των μερών υπάρχει και επιπλέον προϋπόθεση ότι το τρίτο μέρος θα πρέπει να γνωρίζει, να έχει καταλάβει ότι τα, ε, ότι τα έσοδα αυτά προέρχονται από, το, από εγκληματικές πράξεις και στην 24 ότι η δικαστική αρχή θα πρέπει να παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία αμέσως, όμως στην τροπολογία 25 ε, έρεται αυτή η δυνατότητα μπορεί να καθυστερήσει η διαδικασία και η αποδοτικότητα των δικαστικών αρχών και δεν είναι αυτός ο στόχος της ε, τροπολογίας. Να είμαι σαφής ε, κύριε Πρόεδρε, οι αμφιβολίες μας για αυτές τις τρεις τροπολογίες ε, δεν έχουν ως στόχο την μείωση της αποδοτικότητας οποιασδήποτε νομοθετικής πράξης για τη δίμευση. Απλώς θέλουμε να σας καλέσουμε να είστε επιφυλακτικοί για τέτοια ε, νομικά ευαίσθητα ζητήματα, γιατί μπορεί να υπάρχουν ε, ε, νομικά προβλήματα στην νέα νομοθεσία. Σημείωσα επίσης, κύριε Πρόεδρε, ότι η τροπολογία 5 δεν προτείνεται πλέον και το χαιρετίζουμε αυτό. Η αρμοδιότητα της τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το άρθρο 83 για τη συνθήκη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, περιορίζεται σε ένα κατάλογο αξιόπινων πράξεων. Και έτσι και αυτή η δήμευση θα πρέπει να περιορίζεται σε αυτόν τον κατάλογο των ε, σοβαρών αξιόπινων πράξεων. Ίσως να το μετανιώσουμε αυτό βέβαια, αλλά έτσι έχει η συνθήκη. Ευχαριστώ. Okay, if the presidency would like to make a point. Ευχαριστώ. Να δώσουμε το λόγο τώρα στην ε, Προεδρία. Όχι. Εντάξει, τότε ας ε, περάσουμε στον κατάλογο μελετών. Η κυρία Μπορσελίνο. Grazie Presidente. Πρέπει να πω ότι ακούσαμε πολύ ενδιαφέρον την πρόταση οδηγίε του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Είναι κάτι το οποίο περιμένουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα έχει βάρος και πρέπει να χρησιμεύσει στο κοινό καλό το να δημεύονται τα προϊόντα του οργανωμένου εγκλήματος δεν είναι μόνο εξασθένηση της ίδιας εγκληματικότητας αλλά είναι μια επιπλέον εγγύηση για μια κοινότητα πολιτών η οποία έχει φύγει και έχει πέσει θύμα κλοπής και αποδυνάμωσης κάτι το πολύ σημαντικό ιδιαίτερα στην περίοδο την οποία βιώνουμε. Θετικά εκτιμώ λοιπόν την έκθεση της κυρίας Μακοβέη και τη σημερίζομαι εν πολλής. Μου φάνηκε ότι είναι και αρκετά θαραλέα. Με ποια έννοια θέλεις να επιταχύνει και να απλοποιήσει ένα ιδιαίτερα περίπλοκο θέμα για να καταστήσει ξεκάθαρη την εφαρμογή του στην περίπτωση που το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φαινόταν σχετικά θολό και αργό, για συγκεκριμένους λόγους βέβαια αλλά έχει σημασία σε ένα τέτοιο τομέα να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και οι ρυθμίσεις ή νομικές που προτείνονται μπορεί να είναι, πρέπει να είναι εφαρμόσιμες με ξεκάθαρο τρόπο. Και όσο περισσότερες τροπολογίες κατατεθούν, τόσες ε, κερκόπορτες ανοίγονται για να αποδυναμωθεί η πρόταση. Λοιπόν, ε, έχω καταθέσει μια τροπολογία για την ενίσχυση της έκθεσης αυτή τη φορά και επαναλαμβάνω ότι γενικά υποστηρίζω τις απόψεις οι οποίες εκφράστηκαν περιορίζοντας τον αριθμό των εγκληματικών πράξεων σύμφωνα με τη, με νομική βάση. Ένας τόσο πάντως περιορισμένος κατάλογος ενοποιημένα, ε, ενοποιημένες εγκληματικές ενέργειες είναι κάτι το οποίο ε, μοιάζει πάρα πολύ με το λεγόμενο αδίκημα. Το αδίκημα είναι κάτι το οποίο τιμωρείται ε, με μέγιστη ποινή τους 12 μήνες. Είναι προφανές λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχουν όρια έτσι ώστε να μην κατατεθούν τέτοιου είδους, να μην γίνουν δεκτές τέτοιου είδους τροπολογίες. Η κυρία Μακοβέη αναφέρθηκε και σε άλλες τροπολογίες τις οποίες θα αποσύρει είπε, αλλά θεωρώ εγώ ότι το 12, 13 και 14 διευρύνουν το πεδίο κατασχέσεων και περιορίζουν τις δυνατότητες παραγραφής και bis in Μου φαίνεται λοιπόν ότι 9, 10, 15, 16 και 17 είναι σημαντικές τροπολογίες γιατί συγκεντρώνουν σε ένα μοναδικό άρθρο και τις κατασχέσεις που βασίζονται σε καταδίκη και τις κατασχέσεις που δεν βασίζονται σε καταδίκη με δικαστική απόφαση μειώνοντας τις δυνατότητες συνέχισης της δικαστικής διαδικασίας μετά από θάνατο, ασθένεια ή φυγή του κατηγορουμένου. Θα ήθελα να προσθέσω και κάποια άλλη πρόθεση, να προσθέσουμε την δυνατότητα διευρυμένης κατάσχεσης στην περίπτωση κατά την οποία έχουμε να κάνουμε με ποσά τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ τις προσδοκίες που μπορεί να έχει αυτός ο οποίος είναι υποκαταδίκη και ανάλογα και με την κοινωνική επικινδυνότητα του κατηγορουμένου, κάτι το οποίο υπάρχει σε διάφορες χώρες και κάτι το οποίο νομίζω θα μπορέσει να τεκμηριώσει τις εγγυήσει όπου, ε, όπου ε, δεν υπάρχουν, όπου ελείπουν. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και στις κατασχέσεις ε, όχι μόνο στα προϊόντα του εγκλήματος αλλά και στα μέσα του αδικήματος. Σχετικά τώρα με όλα αυτά έχει σημασία όλα αυτά έχουν σημασία όχι μόνο για συμβολικούς λόγους, όχι μόνο για δεοντολογικούς λόγους, αλλά γιατί τα αγαθά που ανήκουν στην κοινότητα των πολιτών Πρέπει να επιστρέψουν σε αυτή την κοινότητα και να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για κοινωνικούς λόγους. Κάτι τέτοιο υπάρχει στην Ιταλική νομοθεσία και είναι κάτι το οποίο έχει δώσει πολύ σημαντικά αποτελέσματα στα όρια βέβαια και, στους με τους περιορισμούς οι οποίοι έχουν παρουσιαστεί και οι οποίοι πρέπει να διορθωθούν μέσω ρυθμίσεων από στο εσωτερικό των κρατών μελών να φύγουν οι περιορισμοί σχετικά με τη χρήση των κατασκευμένων προϊόντων και να περιορίζεται η καταστροφή των προϊόντων μόνο στην περίπτωση που το κόστος της μεταφοράς και χρήσης είναι υψηλότερο από το κόστος καταστροφής. Πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κατάσχεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης και κανόνες δικαστικής συνεργασίας και στον ανακριτικό τομέα. Λόγω του περιορισμένου της νομικής βάσης κάτι τέτοιο δεν θα είναι εφικτό. Θα ήθελα όμως να κατανοήσω την επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει να καλύψει το κενό αυτό γρήγορα, ιδιαίτερα για τις δυνατότητες δικαστικής συνεργασίας και συνεργασίας σε ανακριτικό επίπεδο πριν από κατασχέσεις, από διαδικασίες κατασχέσεων. Νομίζω ότι έχει σημασία και πρέπει η Επιτροπή να προχωρήσει. Ένα σχόλιο προσωπικό εδώ. Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να σέβεται κανείς φυσικά τις εγγυήσει και τα δικαιώματα αυτών οι οποίοι έχουν προβεί στην τέλεση του αδικήματος και οι οποίοι διώκονται δύο. Αλλά μην ξεχνάμε ποτέ ότι ε, πολύ περισσότερο ε, θα πρέπει εξίσου ή πολύ περισσότερο να υπερασπιστούμε και τα δίκαια αυτών οι οποίοι αναγκάστηκαν να πτωχεύσουν λόγω του συγκεκριμένου αδικήματος. Ευχαριστώ κυρία Μπορσέλινο. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την πρότασή της και ιδίως να συγχαρώ την κυρία Μακοβάη για το εξαιρετικό της έργο που εμένα μου δίνει πλήρη ικανοποίηση. Επίσης και όπως και η κυρία Μποσαλίνο, εκφράζω τη λύπη μου και ίσως η κυρία Μακοβέη θα μπορούσε ίσως να επανέλθει για το γεγονός ότι ακύρωσε μια σειρά από τροπολογίες. Εμείς έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία στην Επιτροπή αυτή όπως γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε για όλα τα θέματα οργανωμένου εγκλήματος, διαφθοράς, λεύκανσης χρημάτων. Γι' αυτό δημιουργήσαμε και την Επιτροπή Ειδική για την Εξέταση των Εγκληματικών Ενεργειών η κυρία Αλφανό είναι πρόεδρος και η κυρία Μπορσαλίνο είναι εξέχον μέλο αυτή τη Επιτροπής, όπως και η κυρία Μακοβέη και άλλοι. Και αναμένουμε με μεγάλη αδειμονία την πρόταση αυτή της Κομισιόν. Ξέρουμε ότι οι μαφιόζοι εργάζονται με στόχο το κέρδος και γι' αυτό για τις δικαστικές αρχές και τις διοκτικές αρχές ο στόχος θα πρέπει να είναι η κατάσχεση των αγαθών τους και γι' αυτό αυτή η πρόταση την οποία έχει ζητήσει επανειλημμένα το Κοινοβούλιο είναι να υπάρξει η κατάσχεση ή το πάγωμα των στοιχείων ενεργητικών του των ατόμων αυτών. Λέτε κυρία Κοβέη ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν συνάδουν με την νομοθεσία. Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε ένα άτολμο κείμενο γιατί να μην θέσουμε το ερώτημα στο, στο, νομική, στο νομικό σύμβολο του Κοινοβουλίου ή και της Κομισιόν λέτε ότι η κατάσταση αγαθών τα οποία έχουν δοθεί σε, τρίτου, τρίτους θα πρέπει να συνοδεύεται από κάποια <clears throat> επιφυλακτικότητα όταν όμως κάποιος δίνει ένα διαμέσμα παραδείγματος χάρη σε τιμή πολύ χαμηλότερη από την τιμή αγοράς του αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πρόδειλο. Δεν πρέπει να θεωρείτε ότι οι διοκτικέ αρχέ και οι εισαγγελεί είναι βλάκε, ε, κυρία Μακοβέη. Νομίζω λοιπόν ότι το να σεβαστούμε και τα δικαιώματα των θυμάτων είναι πιο σημαντικό παρά να σεβαστούμε τα δικαιώματα των τρίτων οι οποίοι εμπλέκονται σε τέτοιες συναλλαγές. Εγώ δίνω, εν πάση περιπτώσει, κάθε την απόλυτη μου εμπιστοσύνη προς την κυρία Μακοβέ για να παραμείνει στη θαραλέα γραμμή της και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και στην Επιτροπή ΚΡΙΜ. Εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Αν έχουμε νομικές αμφιβολίες θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα στο νομικό συμβουλό του Κοινοβουλίου. Αλλά κάθε, σας εύχομαι κάθε επιτυχία και πολύ θάρρος σε αυτό το δύσκολο χέρμα. Η κυρία Αλφάνο έχει το λόγο. Και εγώ δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία είπε η Μπορσελίνο και η Ματιό, τις οποίες ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τη Μόνικα γιατί έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά και στον τομέα της κατάσχεσης και στον τομέα της εκ νέου ή μη χρήση από πλευράς των εγκληματιών των αγαθών προϊόντων κλοπής ή απάτης. Θα πρέπει να μην υπαναχωρήσεις όμως Μόνικα, γιατί εμείς σε στηρίζουμε. Αυτό που είπε η Ρίτα Μποσελίνο για μένα είναι κάτι το πολύ συνηθισμένο και ε, θα έλεγα δεν μπορεί κανείς ε, να μην το κάνει δεκτό. Θα πρέπει εμείς σαν κοινοβούλιο πρέπει να κάνουμε μεγάλα βήματα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι τα προβλήματα και ποιο είναι το μέγεθός τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει κάποια σημαντικά βήματα στα πλαίσια του προγραμματός της και κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας το Συμβούλιο είχε εκφραστεί με ξεκάθαρο τρόπο, αλλά δεν θα πρέπει να κάνουμε βήματα προς τα πίσω. Εγώ από την Επιτροπή άκουσα δύο αντιφατικά πράγματα. Πρώτον ότι έχουμε καθυστερήσει και αυτό έπρεπε να το έχουμε ζητήσει εδώ και καιρό και από την άλλη όμως θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηρή σε σχέση με τις νομικές εγγυήσεις και ρυθμίσεις που παρέχει η ε, πρότασή μας και πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Λοιπόν, εμείς έχουμε χάσει δεκαετίες στον τομέα αυτό και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το οργανωμένο έγκλημα συνέχισε και συνεχίζει αυτή τη στιγμή να σωρεύει πλούτο που δεν είναι πλούτος που ανήκει σε συγκεκριμένους πολίτες είναι πλούτος που ανήκει σε 17 κρατημέλη, είναι πλούτος που ανήκει σε 500 εκατομμύρια πολίτες. Γι' αυτό λοιπόν ε, ε, θα ήθελα να ζητήσω ε, Μονίκα να λάβει υπόψη αυτό το οποίο είπε η Ματιέ. Το οργανωμένο έγκλημα και οι μαφιόζικες θα έλεγα οργανώσεις ε, είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένες όταν εμεί κάνουμε κάποιες προτάσεις και τελικά δεν τις θέτουμε σε λειτουργία. Θα ήθελα τώρα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πέρα από αυτά τα οποία είπα, να εκφράσω δύο συγκεκριμένα σημεία απογοήτευσης. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό το οποίο λείπει, είναι μια μορφή καταγγελίας αν θέλετε ή μάλλον μια υπαναχώρηση αρνήθηκε να προχωρήσει με ένα κανονισμό για αμοιβαία αναγνώριση των ενταλμάτων κατάσχεσης. Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μας πει πότε θα καταθέσει αυτή την πρόταση. Και επίσης ελείπουν και οι κανόνες σχετικά με τον προορισμό και την διαχείριση των προϊόντων εγκλήματος. Είναι σαφές λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να εμείνει στα θέματα αυτά τα οποία θεωρούμε βασικά. Σαν πρόεδρος της ΚΡΙΜ και μαζί με τους Σκιώδης θα προσπαθήσω να προχωρήσουμε στη διαδικασία, να τροπολογήσουμε το κείμενο αυτό και η διαδικασία κατάσχεσης της περιουσίας των εγκληματιών αυτή τη στιγμή εντοπίζονται μέχρι τη στιγμή που δημεύονται θα πρέπει να είναι κάτι το ενιαίο ε, ε, και χωρίς προβλήματα και με μεγάλη ταχύτητα σε όλες τις χώρες. Η Επιτροπή είπε ότι η τροπολογία 4 είναι ιδιαίτερα υπερβολική και ότι η τρίτη συνήθως είναι καλή την πίστη. Εγώ δεν έχω γνωρίσει κανένα τρίτο μέρος ε, το οποίο να είναι πράγματι να λειτουργεί καλή την πίστη. Νομίζω ότι οι ανακριτικές αρχές και οι αστυνομικές αρχές μας αποδεικνύουν σε καθημερινή βάση τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε η Ρίτα, γιατί όλες οι εγγυήσει φυσικά για τους κατηγορουμένους, όλα τα δικαιώματα των κατηγορουμένων ε, πρέπει να γίνονται αντικείμενο εγγύησης, αλλά να μην ξεχνάμε ότι κυρίως και θεμελιωδώς αυτό το οποίο πρέπει να σεβαστούμε είναι τα δικαιώματα των θυμάτων. Ευχαριστώ κύριε Αλφάνο. Σας παρακαλώ όλους να έχετε υπόψη σας τους χρονικούς περιορισμούς. Είχαμε προβλέψει μισή ώρα για το συγκεκριμένο σημείο και θα πρέπει να υποδεχθούμε και τον εκπρόσωπο της Ευρωπόλα ο κύριος Ντε έχει στήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ομολογώ ότι η σημερινή συζήτηση δεν με ικανοποιεί και κατανοώ τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχω να αποβάλω αρκετά ερωτήματα, ελπίζω να με προσέχουν. Κατανοώ λοιπόν τη θέση της, Επιτροπ... της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επειδή η Επιτροπή μας, η στο παρελθόν έχει ε, ζητήσει να τηρηθούν δύο αρχές, της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, που ε, γράφονται και στην συνθήκη, οπομένως είναι ευσολογικό. Η Επιτροπή το έκανε αυτό λοιπόν. Αν διαβάσω την έκθεση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το θέμα της επικουρικότητας έχει τύχει λεπτομερούς εξέτασης, ακούσαμε πολλές πληροφορίες το πρώτο ερώτημά μου λοιπόν προς την ε, Κομισιόν είναι ότι θέλω ε, να κατανοήσω το σύνδεσμο με την ε, αξιολόγηση αντικτύπου. Και εκεί πέρα μας παραπέμπουν σε έναν άλλον ιστότοπο, όμως δεν συνδέεται με, τον, με την αξιολόγηση αντικτύπου. Μπορείτε λοιπόν να μου τη στείλετε το συντομότερο δυνατόν, σας παρακαλώ. Μετά για την αρχή της αναλογικότητας η Επιτροπή και πάλι λεπτομερώς εξηγεί γιατί έχει προτείνει κάποια πράγματα και γιατί δεν προτείνει άλλα που ζητούν οι συνάδελφοι της Επιτροπής μου. Και εδώ αναφέρεστε στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπινών Δικαιωμάτων. Εκτός από μία υπόθεση όμως νομίζω δεν έχουμε ε, ένα σύνολο αποφάσεων. και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί Βεβαίω και ε, θέλουμε να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Ταυτόχρονα όμως αυτή τη στιγμή έχουμε τέτοιες μεγάλες προτάσεις της συζυγήτριας, ιδιαίτερα φιλόδοξες και είναι δύσκολο να κατανοήσουμε αν όλες αυτές οι προτάσεις ε, ε, βρίσκονται στην εμβέλεια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ε, έλαβε την εισηγήτρια μία υπόθεση, αλλά εκεί ήταν συγκεκριμένη υπόθεση όπου τα προϊόντα θα χρησιμοποιούνταν για ένα άλλο έγκλημα και εκεί πράγματι η απόφαση έλεγε ότι ε, εφόσον υπάρχει τέτοιο κίνδυνο, επιτρέπεται η δέσμευση και δίμευση. Αυτό είναι συγκεκριμένο όμω για μα. Είναι πολύ δύσκολο όμω να κατανοήσουμε αν βρισκόμαστε εντό του πεδίου των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και θα ήθελα η Επιτροπή να μα δώσει αυτέ τι ε, αποφάσει. Η δεύτερη παρατήρησή μου απευθύνεται στους συναδέλφους εδώ. Ε, σημείωσα τη συζήτηση στην συνάντηση των ε, συντονιστών ε, για τη γνωμοδότηση του Οργανισμού Θεμελιδών Δικαιωμάτων, ακριβώς επειδή είναι περίπλοκο το θέμα. Ταυτόχρονα, οι συνάδελφοι Σκιώδης ε, ζητούσαν παραπάνω ζητούν παραπάνω δεν θέλουν μόνο αυτήν την... δεν αναφέρονται μάλλον σε αυτή την ε, γνωμοδότηση των εμπειρογνωμόνων. Τι θέλουμε λοιπόν εδώ. Κάνουμε μια συζήτηση ε, ε εκπροσωπώντας πολιτικές ομάδες ή ως πρόσωπα. αλλιώ μπορούμε να καταλήξουμε σε μια γνωμοδότηση, μια έκθεση που θα ικανοποιεί τους χειώδεις, αλλά όχι τι πολιτικέ ομάδε. Ας μην βιαστούμε λοιπόν, ας είμαστε προσεκτικοί. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η συγγήτρια θέλει να περιορίσει, για παράδειγμα, το, το πεδίο εφαρμογή για το οργανωμένο άγγλυμα, όπω πρότεινε η Επιτροπή, γιατί αυτό είναι ένα από τα σοβαρά ζητήματα. Αν ε, επεκτείνουμε ε, το πεδίο εφαρμογή, τότε χρειαζόμαστε και άλλη εξολόγηση δικτύπου, για να δείχνουμε ότι το νέο πεδίο εφαρμογή ε, συνάδει με την αρχή τη επικουρικότητα. Και δεν έχουμε μια τέτοια εξολόγηση δικτύπου τώρα. Επομένω, θα ήταν καλό να εξετάσουμε με τη βοήθεια της ε, ε, Επιτροπής ε, και με τη βοήθεια του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, να εξετάσουμε λοιπόν αυτές τις δικαστικέ αποφάσει. και έτσι θα βοηθηθεί και η Επιτροπή μα να πάρει μια τέτοια σημαντική απόφαση και να καταλήξουμε σε συνένεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντεγιόγκ. Είδα ότι σηκώσατε το χέρι σα, κυρία Αλφάνο. Θέλετε να προσθέσετε κάτι. Νομίζω ότι στην ουσία η άποψη των σχεδόν εισηγητών δεν έχει ληφθεί υπόψη συγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωση που έχει ζητηθεί η άποψη από τις διάφορες υπηρεσίες κάτι τέτοιο δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτή είναι η άποψη των σκιωδών και όχι η δική μου προσωπικά. Εντάξει. Ο κύριος Βος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι. Και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στην προσέγγιση η οποία έχει ακολουθηθεί εδώ. Είναι η σωστή. Αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να ακολουθήσουμε γενικά. Ξέρουμε ότι ε, η συνάδελφος, η συγγήτρια ε, πραγματικά ενδιαφέρεται πολύ για αυτό το θέμα και αυτό είναι αξιοθαύμαστο. Υπάρχει βέβαια πίεση χρόνου εξαιτία του μεγάλου αριθμού των θεμάτων που πρέπει να παρακολουθούμε στι διαφορετικέ επιτροπέ, δεν κατάφερα να ε, εξετάσω περαιτέρω αυτό το θέμα. Είναι δύο ή τρία θέματα τα οποία θα ήθελα να αναφέρω και τα οποία μπορούμε μετά να τα συζητήσουμε ίσως διμερώς με την εισηγήτρια. Εγώ πάντα είχα την εντύπωση ότι θέλουμε να ρυθμίσουμε κάτι που αφορά το ποινικό δίκαιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί το ποινικό δίκαιο είναι κάτι το οποίο έχει εξελιχθεί με διαφορετικό τρόπο σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Και υπάρχει μια πολυπικιλία στις ρυθμίσεις. Γι' αυτό <clears throat> δεν ξέρω κατά πόσο αυτά προτείνει η κυρία Μακοβέη θα μπορέσει να ενσωματωθεί στη νομική τάξη των κρατών μελών και κατά πόσο συνάδει με αυτές τις νομικές τάξεις. Υπάρχουν επίσης και κάποιες βασικές αρχές τις οποίες έχουμε εισαγάγει και στην έκθεση του κυρίου Ντε και ίσως και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτές οι βασικές αρχές. Καταρχήν θα πρέπει να έχουμε μία στάση επιφυλακτική για ορισμένες αρχές. Καταρχήν, αυτό που αναφέρεται στην, ε, στις τροπολογίες 3, 6 και 12. Η έννοια του ne bis in idem, το ότι δεν δικάζεται κανείς δύο φορές για το ίδιο αδίκημα, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Επίσης υπάρχουν τα όρια, το θέμα της ιδιοκτησίας και των ορίων που τίθονται στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας από τα συντάγματα των κρατών μας μελών. Το θέμα της ε, παραγραφής, το θέμα της ε, ασφάλειας δικαίου, όλα αυτά είναι ζητήματα και αρχές που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Και επίσης η ε, προαίρεση αθωότητος, το γεγονός ότι θεωρείται κανείς αθώος μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τα ζυγίσουμε και να τα σταθμίσουμε στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αν υπάρχουν τώρα κάποιες αμφιβολίες, νομικού χαρακτήρα αμφιβολίες, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ρυθμίσεις οι οποίες παρακάμπτουν αυτές τις ε, αμφιβολίες και θέτουν το νομικό το κράτος δικαίου σε ένα διαφορετικό δρόμο. Εγώ πιστεύω ότι το κράτος δικαίου είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της τάξης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδαμε τι έγινε στη Ρουμανία όπου υπήρξαν αυθαίρετες ενέργειες μέσα στα πλαίσια του, νομικού, του δικαστικού συστήματος. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι διατηρούμε τον πυρήνα του νομικού συστήματος στην Ευρώπη. Κυρία Αντισέβιτς, αν μπορείτε να είστε σύντομοι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι ένας αριθμός από τα κράτη που έχουν εισαγάγει την κατάσχεση χωρίς προηγούμενη δικαστική απόφαση. Θέλω εδώ να τονίσω ότι και η Κροατία έχει εισαγάγει κανόνες για αποτελεσματική χρήση της κατάσχεσης χωρίς δικαστική απόφαση που επιτρέπουν την κατάσχεση στοιχείων ενεργητικού που έχουν μεταφερθεί σε τρίτους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Λίγιο Πρόεδρο. Ευχαριστώ για τη συντομία σας. Τώρα. Κύριε Πρίβε, βλέπω ότι θέλετε να αναφέρετε κάτι σε σχέση με τα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν από του βουλευτέ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομο. Σα ευχαριστώ για όλε τι παρατηρήσει των βουλευτών. Εγώ δεν έχω πει ότι δεν συμφωνούμε με την ανάγκη να κάνουμε προτάσεις, απλώς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. <clears throat> Μιλάμε για ακυρώσεις που αναφέρονται σε άτομα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τύχη καταδίκηση ή είναι τρίτη σε σχέση με το αδίκημα που διαπράχθη. Πρέπει να τονίσω ότι αυτό το θέμα πέραν όλων των άλλων θεμάτων ποινικού δικαίου που έχουμε αντιμετωπίσει εδώ αντιμετωπίσει διαφορετικές παραδόσεις στο ποινικό δίκαιο των κρατών μελών. Σε ορισμένε χώρε είναι αδύνατο ουσιαστικά να υπάρξει κατάσχεση αγαθών χωρί πρώτερη δικαστική απόφαση. <clears throat> Η πρόταση λοιπόν αυτή που υποβάλλεται είναι θαραλέα, αλλά εδώ τα κρατη θα, ακούσουν, ακολουθήσουν τη δική τους γραμμή στο Συμβούλιο. Θα πρέπει όμως να, είναι, είμαστε εν επιγνώση ότι για ορισμένε παραδόσεις ποινικού δικαίου αυτή η πρόταση είναι τελείως επαναστατική, ενώ σε άλλα κράτη-μέλη μπορεί πράγματι να αντανακλά το τωρινό επίπεδο νομοθεσίας που ισχύει στον ποινικό τομέα. Εμείς θεωρούμε το άρθρο 83 της συνθήκης επιτρέπει μόνο την εναρμόνιση ε, ρητών δικαίου σε σχέση με τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο αυτό. Φυσικά αυτό περιλαμβάνει και το οργανωμένο έγκλημα και δεν εμποδίζει τίποτα τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν περισσότερο. Αλλά οποιαδήποτε νομοθεσία η οποία θα θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα δημιουργήσει και προηγούμενη για όλα τα άλλα δικείμενα που δεν καλύπτονται από τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι η πρότασή μας είναι αυτή τη στιγμή ανεπαρκής, γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το θέμα της δικαστικής αμοιβαίας αρρωγής. Είναι ένα άλλο τμήμα βέβαια της Κομισιόν που είναι αρμόδιο για το θέμα αυτό, όχι το δικό μου. Για τον κύριο Ντε θα έχετε την μελέτη αξιολόγηση αξιολόγησης και αντικτύπου το ταχύτερο δυνατό. Εμείς πράγματι θα πρέπει να ελέγξουμε όλες τις πτυχές θεμελιωδών δικαιωμάτων σε σχέση με αυτή την πρόταση μαζί με την νομική μας υπηρεσία και τους εμπλεκόμενους στα θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν ξέρω αν πρέπει πράγματι να ζητήσουμε και την γνώμη του φορέα προστασίας θεμελιωδών ελευθεριών. Αυτό ίσως θα οδηγήσει σε περαιτέρω καθυστέρηση για την αρχή της επικορικότητας. Πάντα την έχουμε υπόψη μας και γνωρίζουμε ότι υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία των κρατών μελών τα πρόκειται για θέματα ποινικού δικαίου και εναρμόνισης. <clears throat> Πράγματι υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική ανάγκη να νομοθετήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το θέμα αυτό και ευχαριστώ τον Πρόεδρο. Κύριε Μακοβέη, εσείς πάλι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Κομισιόν για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση που έλαβε χώρα. Να αναφερθώ και πάλι σε μερικά από τα επίμαχα θέματα. Για την εμβέλεια του νομοθετήματος βλέπω ότι θέλετε να το κρατήσετε ως έχει. Από νομική έποψη, αν αυτό είναι εντάξει, τότε εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά εμεί ξεκινήσαμε τη συζήτηση χθε με την νομική μας υπηρεσία και τουλάχιστον το σημείο κίνηση τη συζήτηση είναι ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο από ό,τι ορίζει το άρθρο 83 των συνδικών. Εάν τώρα δεν υπάρχει τέτοια, άλλη τέτοια δυνατότητα, εγώ δεν έχω πρόβλημα να παραμείνει η εμβέλεια του νομοθετήματο ω έχει. Επίση, ορισμένοι από εσά θα προτιμούσατε να διατηρήσετε τη δυνατότητα να υπάρχουν αστικέ νομικέ διαδικασίε, δικαστικές διαδικασίες για την κατάσχεση. Εγώ το έλεγξα αυτό και είδα από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά. Θα πρέπει να δούμε αν κατά περίπτωση αν αυτό μπορεί να γίνει ή δεν μπορεί να γίνει. Γιατί εκεί τίθεται και το ερώτημα του, της επιχειρηματολογίας που οδήγησε στην καταδίκη ή στην αθώωση. Για το τρίτο σημείο, το σημείο της κατάσχεσης. Πιστεύω ότι όλοι, <clears throat> όλοι αυτοί τουλάχιστον που έλαβαν το λόγο συμφωνούμε και διαφωνούμε με τη θέση της Κομισιόν για το σημείο αυτό και θέλω και πάλι να αναφερθώ στην αιτιολόγηση που έχει η έκθεσή μου όταν πρότεινα να διαγραφούν όλες αυτές οι περιοριστικές συνθήκες οι οποίες εμποδίζουν την κατάσχεση από αγαθών από τρίτους. Είναι σαφές ότι αν πάρει κάποιος ένα περιουσιακό στοιχείο δωρεάν ή το αποκτήσει με μια τιμή που είναι πολύ κάτω από την τιμή αγοράς, υπάρχει εύλογη υποψία σε σχέση με την προέλευση αυτού του περιουσιακού στοιχείου. Δεν χρειάζεται λοιπόν να το ε, αποδείξει και πάλι το κράτος ότι υπάρχει αυτή η υποψία. Επίσης υπάρχουν κράτη-μέλη που υπάρχει διαφορετική διαδικασία. Η βασική αρχή είναι να παρακολουθήσουμε την πορεία των χρημάτων ανεξάρτητα από τα χέρια στα οποία βρίσκεται αυτό το χρήμα. Αν οι τρίτοι οι οποίοι έχουν πάρει τα περιουσιακά στοιχεία δείξουν καλή πίστη, τότε μπορεί να επιληθεί το θέμα αυτό με το να αναφέρουν και αυτοί πώς έχουν αποκτήσει τα αγαθά αυτά. Οπότε δεν είναι το πρόβλημα του κράτους. Το κράτος θέλει απλώς να ανακτήσει τα χρήματα τα οποία προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες αν κάποιος έχει δείξει αφέλεια ή έλλειψη γνώσης και δεν έχει φανταστεί ότι τα περιουσιακά αυτά στοιχεία προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει την οδό των αστικών διαδικασιών και να, να προσφύγει εναντίον αυτών από τους οποίους απέκτησε τα περιουσιακά στοιχεία. Ξέρω ότι συμφωνείτε όλοι και γι' αυτό θέλω να διατηρήσω το κείμενο ως έχει. Τέλος. για τη διαβούλευση με το φορέα προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών, συμφωνώ με την Κομισιόν ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αυτό θα οδηγήσει μονάχα σε καθυστερήσει και επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά ότι εγώ έχω αναδειφίσει την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από απλώς μια άποψη, μια γνώμη που θα μας δώσει ο φορέας <clears throat> αυτός για τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Γι' αυτό το λόγο δεν βλέπω να υπάρχει από χρόνο λόγος να ζητήσουμε αυτή τη γνωμοδότηση. Και επειδή αυτό εμφανίζεται και σε άλλους ε, φακέλους, όταν ζητάμε διαβούλευση από τη μία πλευρά, ε, θα πρέπει να ζητήσουμε και τη διαβούλευση με την άλλη πλευρά, που είναι στην συγκεκριμένη περίπτωση οι διοκτικές αρχές. Δεν υποστηρίζω λοιπόν την αίτηση γνωμοδότηση προ τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, γιατί δεν έχει υπάρξει επαρκή επιχειρηματολογία για το θέμα αυτό. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βασίζεται στην αρχή της νομολογίας. Μία απόφαση αρκεί για να δημιουργήσει προηγούμενο. Πάντα οι κατασχέσεις βασίζονται σε συγκεκριμένα γεγονότα, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Μπορούμε να δούμε τις περιπτώσεις που έχει αποφασιστεί η κατάσχεση και να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Εφόσον αυτό προβλέπεται από την νομοθεσία, και εδώ θα έχουμε μια νομοθεσία, ο κάθε υπόδικος έχει πάντα το δικαίωμα για ε, αρρωγή από συνήγορο στην υπεράσπιση του. Ωραία. Μπορούμε να σταματήσουμε τη συζήτηση προς το παρόν και να περάσουμε στο επόμενο σημείο με 20-21 λεπτά καθυστέρησης. Ίσως μπορούμε να λειτουργήσουμε λίγο πιο γρήγορα ώστε να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Europol εγκαίρως. 23 το σημείο έγγραφο εργασίας της Κομισιόν σε σχέση με την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την προστασία κέριων στοιχείων υποδομής. Τον Ιούνιο του 2012 η Κομισιόν παρουσίασε ένα έγγραφο εργασίας για το θέμα αυτό, την αναθεώρηση του προγράμματος για την προστασία κερίων υποδομών θα μας παρουσιάσει την αναθεώρηση αυτή η Κομισιόν. Ελπίζω να είναι σύντομη παρουσίαση και μετά αν θέλει ο Θεός και είναι κάποια μέλη τα οποία θέλουν να λάβουν το λόγο θα ακολουθήσει η συζήτηση. Δίνω το λόγο λοιπόν στην Κομισιόν από τον κύριο Κρίστιαν Λάουξ. Έχετε το λόγο κύριε Λάουξ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τηλεγραφικά θα ήθελα να σας εξηγήσω τι ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε στα πλαίσια της προστασίας των κρίσιμων υποδομών, τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Πρόκειται για μια σχετικά νέα ιστορία, αν θέλετε, στις δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης Ξεκίνησε το 2006, σαν να λέγαμε προχθές, με το EPSIT, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για Κρίσιμες Υποδομές. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο αποτελείται από διαφορετικούς πυλώνες. Το πρώτο είναι ένα νομοθετικό μέσο και μια οδηγία σχετικά με τον αντοπισμό και προστασία των μεγάλων βασικών υποδομών πέρα από τα εθνικά σύνορα. Έχει τέσσερα επιπλέον μέτρα η πρόταση αυτή. Είναι ένα μέσο πληροφορικό για να ανταλλάσσουν τα κράτη-μέλη πληροφορίες σε σχέση με τις κρίσιμες υποδομένες. Λέγεται C-WIN. Έχουμε ένα ξεχωριστό οικονομικό πρόγραμμα για να υποστηρίξουμε πιλωτικά προγράμματα για κρίσιμες υποδομές Έχουμε επίσης μια εξωτερική διάσταση, έχουμε ένα ζωηρό διάλογο με τον Καναδά και τις Ηνωμένε Πολιτείε και το πρόγραμμα τέλος προσπαθεί να αναπτύξει την, ε, τη δυνατότητα οι πολίτες να συνειδητοποιούν σωστά τη σημασία που έχει η προστασία των υποδομών αυτών. Εφαρμόζεται το πρόγραμμα αυτό το ΕΨΙΤ εδώ και έξι χρόνια και ήρθε ο χρόνος αναθεώρησης. Η αναθεώρηση νομικά αφορά μόνο την οδηγία, αλλά de facto ασχολείται η, θα έλεγα, μεταρρύθμιση με το σύνολο του προγράμματος. Συνοπτικά, η αξιολόγηση και όλα αυτά τεκμηριώνονται στο έγγραφο που δημοσιεύτηκε τον μήνα Ιούνιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει, εν πάση περιπτώσει, ότι η οδηγία μέχρι τώρα δεν έχει, ε, θα έλεγα, ωφελήσει όσο προβλέπετε. Κοιτάξτε λίγη ησυχία παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζουμε λοιπόν ότι η οδηγία δεν ωφέλησε όσο θα έπρεπε, περιορίζεται μόνο σε δύο τομείς. Τα διαφορετικά κριτήρια και ο τρόπος λειτουργίας της οδηγίας οδήγησε τα κράτη-μέλη να ασχολούνται μόνο με τα θέματα των εθνικών υποδομών, των οποίων θα έλεγα η κατάρρευση ή η καταστροφή θα επηρέαζε και τους γείτονες. Είναι λίγο παράλογο αυτό γιατί μόνο 14 τέτοιες υποδομές εντοπίστηκαν και χαρακτηρίστηκαν έτσι. Μόνο 14 στον τομέα της ενέργειας και στον τομέα των μεταφορών. Ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι η κρισιμότητα ορισμένων υποδομών επηρεάζουν τον τομέα της υγείας, τον τομέα της οικονομίας, στην περίπτωση που υπάρξει μια συνολική διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, τότε τα προβλήματα θα είναι σημαντικά για τη διαχείριση των μεταφορών, για τα χρηματοπιστωτικά κτλ. Φοβάμαι λοιπόν ότι δεν τα έχουμε καταφέρει καλά. Άλλα τμήματα του προγράμματος ήταν σχετικά χρήσιμα. Ο τακτικός διάλογος που έχουμε με τον Καναδά και τη ΣΥΠΑ είναι θετικός ανταλλάσσουμε βέλτιστες πρακτικές και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού και θα δημιουργήσουμε ένα σύνολο μέσων λοιπόν έστω και ε, με ε, την απόσταση του Ατλαντικού και με συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα έχουμε να μάθουμε πολλά ε, από τις εμπειρίες των άλλων το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Επιτροπής δεν δαπάνησε όλα τις δυνατότητες που είχε, το πρόγραμμα SIPS. Θα βρείτε τα παραδείγματα και τις λεπτομέρειες στο έγγραφο. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάναμε μέχρι τώρα και η αξιολόγηση που μπορεί να κάνει κανείς για το EFSIT. Το πρόγραμμα μπορεί να γίνει αντικείμενο ανηθεώρησης επανεξέτασης και θα κάνουμε κάποιες συνολικότερες προτάσεις στις αρχές του 2013. Το πρόγραμμα όπως είπα λοιπόν θα επανεξεταστεί, κάποια μέτρα πρέπει να αλλάξουν ή να απορριφθούν, αλλά βασικός στόχος μας είναι η προστασία των ζωτικών υποδομών μας από κινδύνους δυσλειτουργίας και καταστροφής. Η λογική μας τώρα, και αυτή είναι αν θέλετε μια μορφή ενημέρωσης η ένα θέμα το οποίο συνεχίζεται η επεξεργασία του, προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας λοιπόν στους εξής τομεί. Θέλουμε εμείς ε, η προσπάθεια εντοπισμού των κρισίμων υποδομών να περάσουν σε ένα διαφορετικό επίπεδο την αξιολόγηση των κινδύνων που υπάρχουν στον τομέα των υποδομών στην Ευρώπη. Να περάσουμε δηλαδή από έναν τομεακό θα έλεγα τρόπο εντοπισμού σε έναν ευρύτερο τρόπο πιο οριζόντιο. Αν υπάρξει μια πτώση των πληροφορικών συστημάτων σε ένα νοσοκομείο ή στις μεταφορές ή στον τομέα της ενέργειας, αυτό είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει το σύνολο της υπήρου μας. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι, ποιοι είναι οι κρίσιμοι και να αξιολογηθούν οι τομείς αυτοί και να αξιολογηθούν επίσης οι μορφές διαχείρισης των κινδύνων μέσα σε αυτούς τους κρίσιμους τομείς και πώς μπορούμε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις. Αυτό είναι το πρώτο, το δεύτερο μάλλον ε, βήμα. Ε, το τρίτον, εδώ μπορούμε να κάνουμε κάποια μέτρα παρασκευή συλλογικά για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασκήσεις εκπαίδευσης, ασκήσεις που βασίζονται σε συγκεκριμένα σενάρια, σε επίπεδο περιφερειακό και υποπεριφερειακό και τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη αν ας πούμε δεν τα καταφέρουμε σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο. Τι μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη επιπλέον και εδώ συνεργαζόμαστε με τους εκπροσώπους της ΕΚΟ, έχουν κάποια θα έλεγα κάποιες δυνατότητες ε, παρέμβαση τις επόμενες εβδομάδες μετά από μια μεγάλη καταστροφή στην περίπτωση που υπάρξει μια τέτοια καταστροφή. Τέλος, για τα νομικό κομμάτι. Το πρόγραμμα ΕΨΙΤ ήδη από το 2006 είχε γίνει δεκτό ομόφωνα επί τη βάση του τέος άρθρου 308 που έγινε τώρα 352. Η συνθήκη της Λισαβόνας λοιπόν το άλλαξε αυτό. Έχουμε το 196 το οποίο ασχολείται με θέματα προστασίας του πολίτη και το θέμα δεν είναι η εναρμόνιση νομοθετική των νομικών πλαισίων αλλά το συγκεκριμένο άρθρο ανοίγει την δυνατότητα για μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα και μια ευρωπαϊκή συνεργασία ανάμεσα στις τοπικές και ευρωπαϊκές αρχές έτσι ώστε να υπάρξει ένα ευρύ πεδίο προστασίας. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι θα κάνουμε σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα. Ευχαριστώ την Επιτροπή για το πρόγραμμα εργασίας. Τώρα, αν υπάρχουν παρατηρήσεις... Υπάρχει κάποιο μέλος που θέλει να πάρει τον λόγο. Όχι. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας, λοιπόν. Σας right away the chance to catch up. Επομένως, εξοικονομήσαμε λίγο χρόνο από αυτό το σημείο. Μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 24 για την Europol το πρόγραμμα εργασίας, αξιολόγηση και έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Και να καλωσορίσουμε τον ε, Διευθυντή της Europol. Good to, good to have you here, Mr. Wainwright. We thank you for being here. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Wainwright. Χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ ανάμεσά μας. Ε, ξέρουμε ότι η Επιτροπή μας στους επόμενους μήνες ε, θα παρουσιάσει μια πρόταση για τη Europol που βλέπετε ότι θα είναι ένα από τα ε, σημεία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για τα εσωτερικά ζητήματα. Περιμένουμε λοιπόν αυτή την πρόταση και Μέχρι τότε συνεχίζεται ένας διάλογος. Ο διευθυντής της Europol, κ. Ράιτ, για τα επόμενα 15 λεπτά περίπου θα μας παρουσιάσει τα τελευταία έγγραφα που φορούν την Europol, το πρόγραμμα εργασίας του 2013, η εξωτερική ε, αξιολόγηση και μεθοδολογία. Μετά την παρουσίαση ε, θα δώσουμε το λόγο και πάλι στον κύριο Πρίβε ως ε, διευθυντής Εσωτερικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την κατάσταση για την πρόταση για των Ευρωπαίων και το νέο κέντρο καταπολέμησης ε, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Ας δώσουμε λοιπόν το λόγο στον κύριο Wainwright. Για τα επόμενα 15 λεπτά, μετά βεβαίως θα υπάρξει συζήτηση.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 course, Κύριε πρόεδρε. έχετε Ευχαριστώ κύριε Περιμένουμε να εμφανιστεί η παρουσίαση ισχυρού σημείου μου στην οθόνη. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρουσιάσεις προς τον. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και όλα τα μέλη τη Επιτροπή για την πρόσκληση να σα δώσω ορισμένε γενικέ κατευθύνσει σε σχέση με τι τελευταίε εξελίξει στην Ευρωπόλ που πιστεύω ότι θα πρέπει να ενδιαφέρουν την Επιτροπή σα σε σχέση με τον νέο κανονισμό τη Ευρωπόλ που επίκειται η εξέτασή του και επίση σε σχέση με άλλε εξελίξει οι οποίε είναι πολύ σημαντικέ για την Ευρωπόλ αυτή τη στιγμή συμπεριλαμβανόμενε, όπω όπως είπε και ο πρόεδρο, τη ε, πρόταση για τη δημιουργία ενός κέντρου για την αντιμετώπιση του εγκλήματος. Θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένους στρατηγικούς στόχους που έχουμε θεσπίσει για το πρόγραμμα εργασίας μας το 2013 και επίσης να αναφερθώ και σε ορισμένα άλλα σημεία. Τα μέλη της Επιτροπής σας έχουν προσκληθεί να επισκεφθούν την Ευρωπόλ στο νέο αρχηγείο μας στην Χάγη. Το Νοέμβριο θα γίνει αυτό. Ελπίζω ότι πολλοί από εσά θα χρησιμοποιήσετε αυτή την ευκαιρία μια πολύ καλή ευκαιρία να γνωρίσετε καλύτερα και το έργο μας. Όπως ξέρετε, η Ευρωπόλ υποστηρίζει τις ευρωπαϊκές διοκτικές αρχές και αποτελεί και μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή και αξιολόγηση ε, πληροφοριών σε σχέση με εγκληματικέ ενέργειες με στόχο να είναι ασφαλέστερη η Ευρώπη για όλους τους πολίτες. Όλο και πιο πολύπλοκο και πιο απαιτητικό είναι το περιβάλλον στο οποίο πρέπει να ε, ασκούμε αυτό το λειτουργήμα. Υπάρχουν όλο και περισσότερες αιτήσει για τις υπηρεσίες της Ευρωπόλ, αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης έχουμε σταθερούς ή και μειούμενους πόρους. Η αντιμετώπιση λοιπόν σε καιρούς ε, χαλεπούς οικονομικά του εγκλήματος και της ε, τρομοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ο στόχος της Ευρωπόλ και γι' αυτό μας ενδιαφέρει να μπορούμε να έχουμε ένα πιο αποτελεσματικό οργανισμό ο οποίος να έχει και σαν στόχο να είναι πιο αποδοτικός στις χέριες λειτουργίες του. Το πρόγραμμα εργασίας μας λοιπόν για το 2013 θεσπίζει ένα πλαίσιο με στο οποίο εμείς ελπίζουμε ότι μπορούμε να δώσουμε ένα πιο σημαντικό προϊόν στην Ευρώπη και σημαντικές υπηρεσίες αστυνομικού χαρακτήρα. Ανέφερα την πολυπλοκότητα του πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργούμε. Αναφέρθηκα και στην Επιτροπή σας και στην Επιτροπή ΚΡΙΜ σε σχέση με τις νέες ε, εκφάνσεις του οργανωμένου εγκλήματος, τον τρόπο με τον οποίο είναι όλο και πιο παγκοσμιοποιημένο, ότι έχουν πιο δυναμικό χαρακτήρα σε επιχειρηματικό επίπεδο οι αποδιόμενοι στο οργανωμένο έγκλημα, είναι πολύ πιο ευέλικτοι, κινούνται καλύτερα μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επενδύουν σε πολλές μορφές εγκληματικών ενεργειών και αναμειγνύουν με επιτυχία τις νόμιμες με τις παράνομες δραστηριότητες. Βλέπουμε επίσης να ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα. Πολλές φορές οργανώσεις εγκληματικές από την ε, Δυτική Αφρική χρησιμοποιούν ως ε, αγγελιοφόρους κατά κάποιο τρόπο μέσα εισαγωγικά και ως μεταφορείς ε, εγκληματικές οργανώσεις της Ανατολικής Ευρώπης προς την, οι οποίες μεταφέρουν προϊόντα προς την Νότια Αμερική. Βλέπουμε επίσης να είναι και ένας από τους σημαντικούς χώρους εκδήλωσης οργανωμένη εγκλήματος η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Έχω τώρα τις διαφάνειες αυτές στην ε, ε, οθόνη. Πολλές από αυτές προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα τα αριθμητικά στοιχεία και γι' αυτό είμαι επιφυλακτικός λίγα και αυτά τα στοιχεία. Εγώ λυπάμαι που δεν έχουμε καλύτερες ε, καλύτερα στοιχεία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να κάνουν περισσότερο οι εθνικές αρχές και οι ιδιοκτικές αρχές για να καταλάβουμε καλύτερα το χαρακτήρα του κυβερνοεγκλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά βλέπουμε προς στιγμή ότι είναι πάρα πολλά λεφτά και σίγουρα αυξάνεται ο τζίρος του κυβερνοεγκλήματος κάθε χρόνο. Υπάρχει μια όλο και μεγαλύτερη αίτηση για τις υπηρεσίες της Europol το 2011. Αντιμετωπίσαμε πάνω από από 13.500 διαμεθοριακές υποθέσεις, μια αύξηση 17% σε σχέση με το 2010. Για εφέτος για το 2012 περιμένουμε μια περαιτέρω αύξηση 22%. Μια σημαντική λοιπόν αύξηση στην αίτηση για διοπτικές υπηρεσίες και εφαρμογή του νόμου από τις υπηρεσίες μας. Με άλλο τρόπο μπορείτε να δείτε τα στοιχεία τα οποία λαμβάνουμε στην κύρια βάση δεδομένων μας που εστιάζονται σε 20 περιοχές σχεδίασης. Βλέπετε να υπάρχει μια σημαντική αύξηση των στοιχείων που έρχονται σε μας μεταξύ του 2010 και του 2012. Ουσιαστικά έχουμε σχεδόν τριπλασιάσει τις ε, συμβολές που δεχόμαστε από τα κράτη-μέλη. Όλα αυτά σημαίνουν μεγαλύτερο όγκο εργασίας και μεγαλύτερο όγκο πληροφορίας που πρέπει να διαχειριστούμε και να αναλύσουμε, ενώ συγχρόνω δεν έχει αυξηθεί ο αριθμό των αναλυτών που χρησιμοποιούμε στην Ευρωπόλ. Η διαχείριση λοιπόν αυτού του όγκου εργασίας έχει απαιτήσει μια πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων μας. Μια άλλη απεικόνηση του όγκου πληροφοριών που έρχεται στην Europol βλέπετε συγχρόνως ότι ο αριθμός των ε, αναλυτών που απασχολούμε αυξάνει και τον αριθμό των ε, ευκαιριών λειτουργικής υποστήριξης που δίνουμε στα κράτη-μέλη, ένας από αυτούς τους μηχανισμούς το λεγόμενο mobile office, το κινητό γραφείο, όπου έρχονται οι εμπειρογνώμονες επιτόπου για να βοηθήσουν τους εθνικούς ανακριτές σε δύσκολες υποθέσεις. Φυσικά δεν έχουν οι ίδιοι εκτελεστικές εξουσίες, είναι σε ε, απλώς παρέχουν αρρωγή σε, στις διοκτικές αρχές των κρατών μελών, αλλά έχουν άμεση επαφή με τη βάση δεδομένων μας και επομένως μπορούν να βοηθήσουν με την εμπειρογνωμοσύνη τους. Από το 2009 λοιπόν μέχρι σήμερα έχει υπάρξει έκρηξη στην υποστήριξη αυτού του είδους. Μία άλλη σημαντική αύξηση είναι η συμμετοχή, στη συμμετοχή της Ευρωπόλης σε κοινέ ομάδες έρευνας και ανακρίσεων. Από τότε που έχει αναπτυχθεί αυτό το στοιχείο νομοθεσία για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματο, βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη και οι ιδιοκτικέ αρχέ των κρατών μερών χρησιμοποιούν τι ικανότητε των κοινών ομάδων έρευνα όλο και περισσότερο και αυτό έχει ξεκινήσει και χάρη στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής και τη χρηματοδότηση που δίνει η Κομισιόν και τις ευκαιρίες υποστήριξης των κοινών ομάδων ανάκρισης και έρευνας και φαίνεται ότι υπάρχει όλο και περισσότερη αίτηση προς την Europol και το Eurojust να υποστηρίξουν τέτοιου είδους ενέργειες. Οι, τα καθήκοντα και οι ευθύνες της Europol έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και αυτό περιλαμβάνει το νέο κύκλο πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 8 προτεραιότητες για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο και εδώ η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπόλ παίζει ένα ιδιαίτερο ρόλο συντονιστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή των λειτουργικών σχεδίων που απορρέουν από αυτές τις προτεραιότητες, αλλά επίσης δίνει και την υποστήριξη και την στρατηγική τεκμηρίωση για όλες αυτές τις ενέργειες που απαιτούν μια τέτοια τεκμηρίωση. Ένα έγγραφο για τις προτεραιότητες αυτές θα παρουσιαστεί του χρόνου το Μάρτιο η αυξανόμενη λοιπόν ανάγκη για ενέργειες, ενώ οι πόροι μας παραμένουν σε σταθερό επίπεδο, όπως γίνεται και με τις περισσότερες διοικητικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και γι' αυτό δεν πρόκειται να διαμαρτυρηθούμε ιδιαίτερα, εκτός από το να πω ότι είναι μια όλο και πιο πιεστική πραγματικότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτό το οποίο κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις είναι το εξής. Προβλέπουμε κάποιες εξοικονομήσεις και αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας και ιδίως να εντάξουμε το έργο μας μέσα στον κύκλο πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία έχουν γίνει δεκτά για το 2013 μεταξύ του Διοικητικού μας Συμβουλίου και της Κομισιόν. Βλέπετε λοιπόν ότι μπορούν να προκύψουν εξοικονομήσεις ξεκινήσαμε μια γενική άσκηση περικοπής εξόδων από το 2011 που θα συνεχιστεί και το 2013. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία νέων στρατηγικών, έχει βελτιωστεί η ροή εργασίας και η διαχείριση ηλεκτρονικών εγγράφων, μείωση κατά 5% του κόστου ταξιδίου, μείωση του κόστους μετάφρασης, βελτιώσεις στην ε, λειτουργικότητα, βελτίωση λειτουργικότητας στην διακυβέρνησή μας, μη μικρότερος αριθμός συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν πέσει από 6 σε 4 και μια γενική διαδικασία αναδιοργάνωσης η οποία έχει σε στόχο να εξασφαλίσει και τη δημιουργία του νέου κέντρου κατά του κυβέρνου εγκλήματος, αλλά και να εισαγάγει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη διαδικασία μας, με τη μείωση των θέσεων διαχείρισης στην Ευρωπόλ κατά περίπου 20%. Συγχρόνως προσπαθούμε να αυξήσουμε την αποδοτικότητα των ροών εργασίας μας, ιδίως λόγω του μεγάλου όγκου πληροφοριών που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε ξεκινήσει μια νέα διαδικασία που επιτρέπει μια καλύτερη ενσωμάτωση των διαδικασιών, μικρότερη αλληλοεπικάλυψη και αύξηση των συνεργειών μεταξύ διαφορετικών τομέων εργασίας. Βλέπουμε όλο και περισσότερες διασυνδέσεις μεταξύ των εγκληματικών ενεργειών, παραγωγή στην λαθρεμπορία ναρκωτικών και λαθρεμπορία ανθρώπων. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε ένα πιο ευέλικτο περιβάλλον για ανάλυση στοιχείων. Αυξημένη στρατηγική συνεργασία με ορισμένου χώρου του ιδιωτικού τομέα. Ιδίω αυτό είναι σημαντικό για ενόψη του έργου μα στο κύβερνο έγκλημα μια αύξηση ικανότητες ανείχνευσης ε, χρηματοοικονομικών συναλλαγών και καλύτερη διαλειτουργικότητα με άλλους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους φορείς όπως η Ιντερπολ. Ο δεύτερος κύριος στόχος μας για το χρόνο επομένως είναι να υποστηρίξουμε τις ε, δραστηριότητες που αντιμετωπίζουν εγκληματικές απειλές μέσα στην ευρωπαϊκή πολιτική. Σας ανέφερα τις 8 προτεραιότητες, τις οποίες γνωρίζετε ήδη. Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι στην Europol, Ευρωπόλ να εστιάσουμε την προσπάθειά μας για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών. Και όπως είπα το 2013 θα κάνουμε προσπάθεια να έχουμε μια συνολική αξιολόγηση των απειλών από το οργανωμένο έγκλημα. Κάποια μέλη της Επιτροπής σας μας έχουν ζητήσει να τους εξηγήσουμε καλύτερα την μεθοδολογία για την νέα σόκτα όπως αναφέρεται. Εμείς έχουμε επενδύσει πολλή προσπάθεια στο να βελτιώσουμε την μεθοδολογία στον τομέα αυτό και να μπορούμε να έχουμε ένα σύνολο συμπερασμάτων που να είναι τεκμηριωμένα στον τομέα αυτό. Η μεθοδολογία της ΣΟΚΤΑ αναφέρεται σε ένα δημόσιο έγγραφο το οποίο έχει συνταχθεί και με τη συμμετοχή εμπειρογνωμών από τα κρατη αλλά και από μελών από τον ακαδημαϊκό χώρο και ο στόχος είναι να αναλύσει το χαρακτήρα και τις απειλές που μπορούν να προκύψουν από ομάδες οργανωμένου εγκλήματος αλλά επίσης και των δραστηριοτήτων τις οποίες διενεργούν. Είναι αυτή η μεθοδολογία, είναι καλύτερη από τις προηγούμενες μεθοδολογίες και θα πρέπει να μας οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης, στο πρόγραμμα εργασίας μας θα αποδώσουμε έμφαση στο να βελτιώσουμε τα συστήματα ανάλυσης, να αναπτύξουμε μια πιο μεγάλη μόνιμη ικανότητα για να δίνουμε καλύτερες αναφορές στα κράτη-μέλη και στις αρχές του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν αναδύονται νέες πηγές απειλών από το οργανωμένο έγκλημα, να αυξήσουμε και τη λειτουργία της ΣΥΕΝΑ του συστήματος ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών. Είναι ένα κέντρο που χρησιμοποιείται, ένα σύστημα που χρησιμοποιείται από τα περισσοτερα κάτι κράτη-μέλη. Για το μέλλον. Και εν ώψη ενός νέου κανονισμού για την Ευρωπόλ, διότι όπως ξέρετε η Κομισιόν έχει ξεκινήσει μια ανεξάρτητη έρευνα του νομικού πλαισίου της Ευρωπόλ που γίνεται από τον οργανισμό RAND. Όλα αυτά γίνονται λοιπόν με στόχο να βελτιώσουν το έργο της Ευρωπόλ και να οδηγήσουν σε μια νέα πρόταση για την Κομισιόν. Ποια είναι τα συμπεράσματα που μπορώ να σας δώσω από αυτή την αξιολόγηση από τον Νίκο Ραντ. Ήδη τον Ιούνιο ε, έχουν δημοσιευτεί τα έγγραφα αυτά, έχουν δοθεί στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και έχετε τουλάχιστον τη σύνοψη αυτή της έκθεσης. Καταρχήν, θεωρούν ότι η αξία της Ευρωπόλ στα κράτη-μέλη είναι όλο και πιο σημαντική στον τομέα της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Αλλά κάνουν κάποιες προτάσεις για να είναι πιο αποτελεσματική η Ευρωπόλ στο μέλλον. Απλώς θα αναφέρω ένα εδίο. ιδίω αυτό το οποίο αφορά το επίπεδο της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπόλ, ότι υπάρχει πολύς χώρος για βελτίωση, υπάρχουν ακόμα τεράστιες ανισομέρειες σε σχέση με τις πληροφορίες που, που συμμερίζονται ορισμένα κράτη μεταξύ τους και με την Ευρωπόλ. Παρά το γεγονός ότι έχουμε βελτιώσει σημαντικά την τεχνική ικανότητα βάσει της οποίας μπορεί να υπάρχει η διάδοση πληροφοριών, βασιζόμαστε σε μεγάλο βαθμό σε μια κουλτούρα στους διοκτικούς οργανισμούς ώστε να εκτιμήσουν καλύτερα την αξία τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πιστεύω ότι ο κανονισμό αυτό στο βαθμό του δυνατού θα πρέπει να λάβει υπόψη την ανάγκη να παροτρύνει καλύτερα επίπεδα ανταλλαγή πληροφοριών στο μέλο. Η ΡΑΝΤ επίση συνιστά ο νέο κανονισμό να δώσει περισσότερε εξουσίε για την υποστήριξη ερευνών σε εγκληματικέ δραστηριότητε και ενδεχομένω να υπάρχει και χρηματοδότηση αυτών των ενεργειών. Αυτό έχει λειτουργήσει πολύ καλά μέχρι στιγμή και έχει καταδειχθεί ότι είναι ένα από τους κέριου τομείς εργασίας μας. Για να έχουμε και μεγαλύτερη ευκαμψία της επεξεργασίας στοιχείων, όταν έχουμε πολύ μεγαλύτερε ροές πληροφοριών, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, σύμφωνα με τη ΡΑΝ τουλάχιστον, στο να ξεπεραστούν οι ορισμοί των χωριστών συστημάτων επεξεργασία. Αυτό είναι ένα τεχνικό κυρίω θέμα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι πιο μεγάλη και η ικανότητά μας όχι μόνο να αναλύουμε τα δεδομένα, αλλά συγχρόνως να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα του συστήματος προστασίας δεδομένων. Ένα τελευταίο σημείο που θέλω να αναφέρω σχετικά αφορά την μελλοντική σχέση της Ευρωπόλ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές τους τρόπους με τους οποίους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να έχει πιο αποτελεσματικό τρόπο να ασκεί τον κοινοβουλευτικό του έλεγχο έναντι της Ευρωπόλ και εγώ προσβλέπω στο να απελάβει ο κανονισμός και τα εργαλεία με τα οποία θα μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο, όπως παραδείγματος χάρη καλύτερη κοινοβουλευτική πρόσβαση στα έγγραφα της ε, Ευρωπόλ, διαβαθμισμένα έγγραφα βάσει μιας ε, διαδικασία που θα θεσπιστεί και έχουμε ήδη συζητήσει με τον κύριο Αγγιλάρ για το θέμα αυτό και θα συνεχίσουμε τις προσπαθίες μας προς τα εκεί. Εν κατακλείδη, κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπόλ, όπως βλέπετε και από τα στοιχεία που σας έχω δώσει, αποκτά όλο και μεγαλύτερη ε, ικανότητα, μεγαλύτερη ένταση στην εργασία της. Παρ' όλα αυτά, το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε περιλαμβάνει όλο και πιο πολλές και πιο πολύπλοκες προκλήσεις Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να εξυγχρονίσουμε τις ικανότητές μας, να κάνουμε πιο αποτελεσματική την εργασία μας, όπως και όλοι οι άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελπίδα μας είναι ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να βασιζόμαστε στην υποστήριξη της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου εν, γέρι, γέννη για να υπάρχουν τα απαραίτητα χρηματοδοτικά και άλλα μέσα προς την Ευρωπόλια για να φέρει σε πέρα στην εντολή της και προσβλέπω στη συζήτηση που θα ακολουθήσει με το Συμβούλιο, την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο για την έγκριση του νέου κανονισμού της Ευρώπη. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Βάινράιτ. Σας ευχαριστούμε για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Μας ενημερώσετε για τις ε, αναμενόμενες εξελίξεις σε ό,τι αφορά αυτόν τον ε, πολύ σημαντικό φορέα στον τομέα της καταπολέμησης ε, του εγκλήματος ε, στην Ευρώπη και της ε, συνεργασίας μεταξύ αστυνομικών αρχών και αρχών επιβολής του νόμου. Τώρα, να δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή. Ο κύριος Πρίβε, εκ μέρου της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, θα ήθελε να κάνει και αυτός μια παρουσίαση και μετά θα, θα δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους. Σίγουρα θα υπάρξει χρόνος για ερωτήσεις και τοποθετήσεις. Κύριε Πρίμπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο για να μπορέσω και εγώ να σας ενημερώσω για το τι συμβαίνει με τον κανονισμό για την Ευρωπόλ. Δεν προτίθεμαι να κάνω παρατηρήσεις ε, στην ε, παρουσίαση του ε, Διευθυντή της Europol για το πρόγραμμα εργασίας του 2013. Όπως είπε και ο ίδιος, εμείς έχουμε στηρίξει πλήρως αυτό το πρόγραμμα εργασίας. Για την επερχόμενη πρόταση κανονισμού για την Europol, πολλά που ήθελα να πω δεν χρειάζεται να τα πω γιατί συμφωνώ απόλυτα με τον Διευθυντή. Εμείς ε, είμαστε διατεθειμένοι να υποβάλουμε αυτή την πρόταση φέτος. Ε, όπως έφερε και ο κύριος Βαϊνβράιτ, είχαμε την ανεξάρτητη μελέτη ε, του ΡΑΝΤ αυτού του οργανισμού που βασίστηκε σε ευρεία διαβούλευση των εμπλεκομένων με συμμετοχή των κρατών μελών, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουμε λοιπόν μια πολύ καλή εικόνα για το τι θα μπορούσε να βελτιωθεί, να αλλάξει και το καθεξής. Και αυτή τη στιγμή στην, ε, στο ιστορικό της Επιτροπής ε, γίνεται η αξιολόγηση αντικτύπου που βεβαίως ε, θα αξιοποιήσει την μελέτη της ΡΑΝΤ ως βάση και στη συνέχεια του έτους θα σας υποβάλουμε πρόταση. Αυτό που είναι σημαντικό σε αυτή την πρόταση είναι ότι θέλουμε να κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις για την ε, βελτίωση της αποδοτικότητας ε, του οργανισμού της Ευρωπόλ και να γίνει μια ευθυγράμμιση με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Όμως, έχουμε έναν φορέα που όπως ξέρετε όλοι εργάζεται ήδη πολύ ε, αποτελεσματικά. Δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη να κάνουμε να διορθώσουμε τη λειτουργία του. Ήδη λειτουργεί πολύ καλά. Η ευθυγράμμιση με την ε, Λισαβόνα της Ευρωπόλ είναι βεβαίως σημαντικό από πλευράς ε, θεσμικής και αυτό συμπεριλαμβάνει ε, την βελτιωμένη κοινοβουλευτική εξέταση και έλεγχο της Ευρωπόλ όπως αναφέρεται στο άρθρο 88 της συνθήκης. Παρεμπιπτόντω, αυτό το άρθρο αναφέρεται και στην ε, λογοδοσία του, της Ευρωπόλ απέναντι ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και αυτό το έχουμε συζητήσει σε αρκετέ συναντήσει. Πρέπει να δούμε πώ ακριβώ θα γίνει αυτό. Ε, Προτείνουμε αυτή η κοινοβουλευτική εποπτεία να επικεντρωθεί στον προπολογισμό, την ε, διαχείριση της πολιτικής και των οικονομικών πόρων και για να, να διασφαλιστεί ο διαχωρισμός των εξουσιών ε, δεν προτείνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια να συμμετάσχουν ε, στην καθημερινή διαχείριση του φορέα. Η ευθυγράμμιση με τη Λισαβόνα της Ευρωπόλου επίσης είναι μια εξαιρετική ε, ευκαιρία για την Ευρωπόλ να διορθώσει κάποιες ελλείψεις, ε, αν θα μπορούσα να τις αποκαλέσω έτσι, όπου θα μπορούσε να καταστεί ακόμα πιο αποδοτικό, αποδοτικός ο φορέας. Τα είπε και ο κύριος Βέινβραϊτ βέβαια αυτά. Πρέπει να υπάρχει μια αυξημένη ετοιμότητα των κρατών μελών να ενημερώνουν την Ευρωπόλ, να συνεργάζονται μαζί της. Ε, εδώ δεν ξέρουμε αν πρόκειται για θέμα αλλαγής ε, του ρυθμιστικού πλαισίου των κανόνων ή ε, αλλαγής της νοοτροπίας σε αστυνομικές αρχές των κρατών μελών. Ίσως να μην είναι και ότι το καλύτερο να ε, ε, επιβάλλουμε κανόνες. Ίσως καλύτερο θα ήταν να ξεκαθαρίσουμε λίγο τους κανόνες, να αλλάξουμε νοοτροπίες και να γνωρίζει ο καθένας ότι αν θέλουν πληροφορίες από την Europol και αυτοί θα πρέπει να ε, συνδράμουν. Επίσης πρέπει να ε, γίνεται ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της Ευρωπόλ και αντίστοιχων οργανισμών τρίτων ε, χωρών και στη τη της Λισαβόνας αναφέρεται ότι δεν θα μπορεί πλέον ε, η Ευρωπόλ να συνάπτει τέτοιες συμφωνίες. Πρέπει να ακολουθείται η συνήθιση διαδικασία των διεθνών συμβάσεων, δηλαδή ε, απόφαση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Είναι λοιπόν δύσκολο αυτό το θέμα. Τώρα για την ανταλλαγή των... Ε, α, ας ξεκινήσω την αρχή μάλλον. Σκεφτόμαστε να προτείνουμε την εισαγωγή δυνατότητας της Ευρωπόλ για ανταλλαγή πληροφοριών με ε, ιδιωτικούς φορείς, το οποίο δεν είναι σίγουρο ακόμα, αλλά σε κάποιους τομείς, ιδιαίτερα του εγκλήματος στην κυβερνοχώρα, αυτό είναι σημαντικό. Βεβαίως υπάρχουν ε, κάποιοι προβληματισμοί ε, σε ό,τι αφορά την προστασία δεδομένων. Η αύξηση της αποδοτικότητας ε, σχετίζεται και με την πιο ευέλικτη διαχείριση πληροφοριών. Η Ευρωπόλ φημίζεται βέβαια για τα υψηλά πρότυπα προστασίας δεδομένων. και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο αυτή την ευελιξία, ε, διατηρώντας όμως το υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, ένα πιο οριζόντιο θέμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την σύνταξη αυτής της πρότασης κανόνες που αφορούν τη διακυβέρνηση, την ε, λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, ε, ο διορισμός του Προέδρου, του Διευθυντή. Ε, η Επιτροπή κατόπιν μακράς συζήτησης με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο βεβαίως και επιθυμεί να υπάρχουν εναρμονισμένοι κανόνες στους πάνω από 30 οργανισμούς πια και θα υπάρχουν προτάσεις και από αυτού. Αυτά είχα να πω προς το παρόν για την ε, πρόταση για κανονισμού για την Ευρωπόλ. Πολύ σύντομα για το Ευρωπαϊκό Κέντρο ε, του Εγκλήματος για τον Κυβερνοχώρο που δεν συνδέεται ε, ευθέως με την πρόταση κανονισμού γιατί πρόκειται για νέο καθήκον της Ευρωπόλ μετά την αναθεώρηση της νομικής βάσης βάσει των προτάσεων της Επιτροπής το Μάρτιο που έτυχαν τη συνένεσή σας ότι δηλαδή η Ευρωπόλ θα διοργανώσει αυτό το κέντρο βάσει των όσων έχουν ήδη κάνει μέχρι τώρα. Ε, οι προετοιμασίες οδεύουν καλώς. Βεβαίως πρέπει να εξετάσουμε ακόμα τις ε, οικονομικές ανάγκες ε, αυτού του κέντρου. Δεν είναι κάτι πιο νέο στοιχείο στην νομική βάση της Ευρωπόλ. Βεβαίως όμως πρόκειται για νέα αρμοδιότητα ε, επί της ουσίας, ότι δηλαδή στην καθημερι... στο καθημερινό τους έργο πρέπει να κάνουν ακόμα κάτι παραπάνω. Και έτσι υπάρχουν και κάποια οικονομικά ζητήματα. Ε, το, μια, τη στιγμή που όλοι οι οργανισμοί, ακόμα και τα κράτη-μέλη, κάνουν περικοπές. Από συζητήσεις με την Ευρωπόλη όμως είμαστε αρκετά αισιόδοξοι. Και θεωρούμε ότι όλα πάνε καλά και θα ε, γίνουν όπως αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση του Μαρτίου της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρίπκε για την περιγραφή της κατάστασης της προτινόμενης λισαβονοποίησης εισαγωγικά της Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και νομίζω ότι σύμφωνα ακριβώ και με το πρόγραμμα δράσης ε, της Στοκόλμης πρέπει να προχωρήσετε. Αυτό προβλέπει έτσι και αλλιώς και η συνθήκη της Λισαβόνας. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να δείξουμε ότι είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε και μπορούμε να λάβουμε ε, υπόψη μας τις πραγματικές ανάγκες για την καταπολέμηση του διεθνικού εγκλήματος. Αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη να προχωρήσουμε με ένα νέο νομικό μέσο, το οποίο θα συμπεριλάβει την Europol στον χώρο Τζάι. Ακούσαμε λοιπόν την παρουσίαση του κυρίου Wainwright Ακούσαμε επίσης και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τώρα τα μέλη της Επιτροπής. Ο κύριος Διέστε Μέρα έχει πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ και για τα λόγια σας που άκουσα με μεγάλη ευχαρίστηση. Θέλω να ευχαριστήσω αυτά που είπε ο, τον Διευθυντή της Ευρωπόλ για την παρουσία του που είναι πάντα χρήσιμη και για αυτά που μας παρουσίασε σε σχέση με το πρόγραμμα εργασίας αυτού του φορέα. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τον κύριο Πρίβε από την Κομισιόν για τις πληροφορίες που μας έδωσε για τον νέο κανονισμό της Ευρωπόλ. Απλώς θέλω να κάνω κάποια σχόλια. Εγώ προτιμώ τα σχόλια από τις ερωτήσεις. Τα σχόλια που κάνω είναι τα εξής. Θα ήθελα το λεγόμενο κινητό γραφείο, το mobile office, να είναι ένα στοιχείο το οποίο να υποστηριχθεί όλο και περισσότερο σε λειτουργικό επίπεδο. Ξέρω, κύριε Διευθυντά, ότι αυτά είναι στοιχειώδη. Ότι για την ε, Ευρωπόλη να πάρει το να έχει όλο και περισσότερες δυνατότητες λόγω των αρμοδιοτήτων που έχει από αποκομίσει και σε σχέση με τη δημιουργία μεικτών ε, υπηρεσιών το Mobile Office είναι ένα πρώτο βήμα. Τώρα, για το σχέδιο που έχετε για το κυβερνό έγκλημα. Μιλήσατε για ένα νέο εγχείρημα, κύριε Πρίβε. Αλλά αυτό είναι ουσιαστικά μια πρόταση της Κομισιόν. Δεν μπορεί να γίνει ένα νέο εγχείρημα χωρίς χρηματοδότηση. Όταν έχουμε ένα νέο και σημαντικό εγχείρημα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω προϋπολογισμός. Δεν μπορούμε λοιπόν απλώς να κάνουμε φραστικές δηλώσεις. Εάν θεωρείται είναι τόσο σημαντικό και τόσο απαραίτητο το νέο αυτό κέντρο για τον αγώνα κατά του κύβερνο εγκλήματος. είναι προφανές ότι θα πρέπει να προβλέψετε και για την απαραίτητη χρηματοδότηση του από τον προϋπολογισμό. Η αξιολόγηση από την ΡΑΝΤ ήταν επίσης πολύ ενδιαφέρουσα και είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης για τον νέο κανονισμό. Εγώ χαίρομαι που λέτε ότι το Νοέμβριο ήδη θα έχουμε μια πρόταση κανονισμού για την Ευρωπόλ, το νέο κανονισμό. Και όπως είπε και ο πρόεδρος μας, η Επιτροπή μας δεσμεύεται για να εργαστεί ώστε να υπάρξει ένα σωστά προσαρμοσμένο στις συνθήκη Λισαβόνας νομικό εργαλείο, ο κανονισμός αυτός. Όπως είπα και για το mobile office, το κινητό γραφείο, Συγχρόνω, χρειάζεται βελτίωση και στην ανταλλαγή πληροφοριών. Θα πρέπει να υπάρξει σημαντική βελτίωση ώστε η Ευρωπόλ να έχει τη δυνατότητα να απολαμβάνει τις απαραίτητες εμπιστοσύνης που κερδίζει μέρα με τη μέρα. Ένα ερώτημα θα θέλω να θέσω στον κύριο Wainwright, γιατί εσείς οι Βρετανοί χρησιμοποιείτε τη γλώσσα σας πολλές φορές με τρόπο ιδιαίτερα επακριβή και άλλες φορές με τρόπο λίγο νεφελώδη. Θέλω μία διευκρίνηση. Όταν λέτε σε σχέση με τις αναλυτικές ικανότητες της Ευρωπόλ να υπάρξει ακύρωση των διαφορών στα συστήματα πληροφόρησης. Τι μιλάμε. Αν μιλάμε για αυτό το οποίο νομίζω εγώ ότι μιλάτε, το υποστηρίζω. Αν μιλάτε όμως για τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος, όπου μπορούν να παρεμβαίνουν και άλλοι φορείς, αν μιλάτε γι' αυτό, αν θέλετε να ε, ακυρωθούν όλες οι διαφορές μέσα στην Ευρωπόλη, τότε είναι διαφορετικό. Τέλος, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στον εαυτό κανονισμό και το λέω σε εσά κύριε Πρίλε στην Κομισιόν γιατί χρησιμοποίησατε μια έκφραση που δεν είναι αυτή η οποία αρέσει στο Κοινοβούλιο. Μιλήσατε για εποπτεία. Εμείς όμως ως Κοινοβούλιο μιλάμε για έλεγχο. Άλλο η εποπτεία, άλλος ο έλεγχος από ένα Κοινοβούλιο. Εμείς στο στον κανονισμό θέλουμε να τονίσουμε την έννοια του ελέγχου και θέλουμε να καθοριστεί τι σημαίνει αυτή η έννοια του ελέγχου. Φυσικά δεν θα επηρεάσει τη διαχείριση σε καθημερινό επίπεδο της Κομισιόν. Αλλά θέλουμε να έχουμε ένα αποτελεσματικό και ισορροπημένο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και αυτό αναφέρεται και στο άρθρο 88 της Συνθήκης της Λισαβόνας, αλλά πρέπει να ονομάζεται έλεγχος και όχι εποπτεία απλώς και παρακολούθηση. Συγχαρητήρια και κάθε επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστώ κύριε Διαστεμέρα. Σας ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα και τον κύριο Wainwright και τον κύριο Πρίμπερ να τους ευχαριστήσω για τις προ... προτάσεις τους. Βέβαια αυτά που είπανε είναι πραγματικά συνοπτικά. Αν δει κανείς το χαρτοβασίλειο το οποίο συνοδεύεται συνοδεύει την νέα πρόταση της Κομισιόν, τις έρευνες και τις μελέτες που έχουν γίνει και δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να τα αναγνώσουν όλα αυτά οι συνάδελφοι. Ο κύριος Ράιτ αναφέρθηκε πολύ καλά στην συνεργασία που λαμβάνει η χώρα με τις εθνικές αρχές και την υποστήριξη που δίνει η Ευρωπόλη σε αυτές τις αρχές. Όλα αυτά είναι πολύ θετικά, αλλά αναφέρθηκε και σε ορισμένα σημεία τα οποία η Επιτροπή, η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να τα συζητήσει πολύ σε βάθος εάν πρόκειται να υπάρξει μια τροποποιημένη σχέση της Ευρωπόλ με τις εθνικές αρχές. Επίσης όταν μιλάτε για το κέντρο, για το κυβερνοέγκλημα, εγώ θα ήθελα να ξέρω τι πιστεύετε ότι πρέπει ένα τέτοιο κέντρο να κάνει και ποιε θα πρέπει να είναι και οι δράσει των κρατών μελών σε αυτό τον τομέα. Και ώστε να μην γίνονται όλα μονάχα σε ένα κεντρικό επίπεδο, θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη σαφήνεια σε σχέση με την κατανομή αρμοδιοτήτων. Εγώ έχω σταθεί όμως ιδιαίτερα και έχω εντυπωσιαστεί με αυτά που λέτε για τη συλλογή δεδομένων. Και ο κύριος Πρίβε και ο κύριος Wainwright αναφέρθηκαν σε ορισμένα σημεία για την χωριστή, τα χωριστά συστήματα επεξεργασίας δεδομένων. Αυτό το έχουμε συζητήσει στην ε, ε, Επιτροπή μας ότι όσο πιο πολλά συστήματα υπάρχουν, τόσο πιο εύκολο είναι να υπάρξουν καταχρηστικές αντιμετωπίσεις. Πρέπει να υπάρξει ευελιξία. Λέτε όμως επίσης και για την παράδοση στοιχείων σε τρίτες χώρες. Σε ποιες χώρες και για ποιες ανάγκες. Η μελέτη RAND αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρχει επεξεργασία και ευαισθητών στοιχείων και αναφέρεστε και σε μια ανταλλαγή στοιχείων σε ιδιωτικούς φορείς. Ποιους φορείς εννοείται και προς ποιο σκοπό. Και εμένα με εντυπωσιάζει επίσης ότι αναφέρεται και επί τη βάση της πρότασης της κυρίας Ρέντινγκ για ένα κανονισμό προστασίας δεδομένων. Υπάρχει ένας κανονισμός για τον δικαστικό τομέα στα θέματα αυτά, αλλά υπάρχουν πολλές ε, χώρες μέλη που δεν θέλουν να προχωρήσουν σε κάποιες διαπραγματεύσεις σε αυτό το σημείο για τα δεδομένα και αυτό το θεωρώ λαθασμένο. Νομίζω ότι αυτό λοιπόν πρέπει να το συζητήσουμε ιδιαίτερα ποιε θα είναι και οι συνέπειες που θα προκύψουν για το σημείο αυτό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητήσουμε όχι μονάχα όταν θα έρθει επιτάπητος ο νέος αυτός κανονισμός, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αντιμετώπιση ευαισθητών δεδομένων από τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων και σε ποιους φορείς μπορούν να δίδονται ε, από την, ε, από την Ευρωπόλ και σε ποιους όχι. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Κύριος Φάινχάουζερ. Σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Πρόεδρε. όπως και ο προ, προλαλής σας, θέτω το θέμα του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και θα ήθελα να ξέρω ποιες είναι και οι προδιαγραφές και οι κανόνες σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων. Εγώ σίγουρα χαίρομαι για το γεγονός ότι έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Ήταν πάρα πολύ θετική η εξέλιξη της Ευρωπόλ και είναι ένα νευραλγικό μέσο για τον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Είπατε βέβαια ότι δεν χρειαζόσαστε περισσότερες αρμοδιότητες, αλλά υποστηρίζετε περισσότερο τη δημιουργία ενός πιο έφορου κλίματος συνεργασίας με τις ε, εθνικές αρχές. Αυτό το βρισκό Και επίσης κάτι το οποίο αναφέρθηκε και προηγουμένως, το ερώτημα είναι τι δημοσιονομικούς πόρους θα, χρησιαστείτε για να μπορέσετε να φέρετε πέρας, σε πέρας το ρόλο σας τη στιγμή που έχετε να αντιμετωπίσει όλο αυξανόμενες απειλές και προκλήσεις. Ποια είναι τα πρόσθετα μέσα του προϋπολογισμού που χρειάζεστε και αυτό θα ήταν ενδιαφέρον να ξέρει και η δική μας Επιτροπή γιατί θα πρέπει στην επόμενη άσκηση του προϋπολογισμού να ενσωματώσουμε αυτά τα χρήματα. Θα ήταν χρήσιμο να έχουμε αυτές τις πληροφορίες λοιπόν η κυρία Χόλμαϊρ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν ότι χαίρομαι για την δυνατότητα να έχουμε αυτές τις πληροφορίες από την πλευρά της Ευρωπόλ εν ώψη του νέου αυτού κανονισμού ο οποίος θα εξεταστεί και σας ευχαριστώ και για τις ε, Λεπτομέρειε που μας έχετε δώσει. Φυσικά δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τον κύριο Wainwright να μας δώσει όλες τις λεπτομεριακέ πληροφορίες οι οποίες ουσιαστικά απαιτούν ώρες συνεδριάσεων με την ε, Ευρωπόλ. Εμείς έχουμε 10-15 λεπτά το πόλι. δεν μπορούμε να τα μάθουμε όλα. Δεν πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε ίσως ε, πάντα καχυποψία σε σχέση με την ε, επεξεργασία δεδομένων γιατί μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη αδικημάτων εάν έχουμε τα αντίστοιχα στοιχεία. Μπορεί δηλαδή ένα κράτος μέλος να παίξει ένα ρόλο βοήθειας για την πρόληψη σε άλλα κράτη-μέλη και εδώ παίζει το ρόλο του διαμεσολαβητή η Ευρωπαϊκή η Ευρωπόλ, συγγνώμη, και σε σχέση με το κυβερνοέγκλημα και την αντιμετώπιση του. Αυτό είναι μια από τι σημαντικότερε αρμοδιότητε που μπορεί να έχει η Ευρωπόλ και θέλω να θέσω σχετικά το ερώτημα στον κύριο Wainwright αν μπορεί να μας πει πώς θα μπορούσε να υπάρξει ένα σύστημα πρόληψης για, την, ε, για τον, που θα εμπόδιζε τα μεγάλα αδικήματα τα οποία μπορούν να λάβουν χώρα στο, στο διαδίκτυο και όχι μοναχά τις μικρές παραβάσεις. Και επίση θα ήθελα να σταθώ και πάλι στο θέμα τη ε, καχυποψία που υπάρχει εναντίον τη Ευρωπόλ ότι θέλει να τα συγκεντρώσει, να συγκεντρώσει όλα στα χέρια της, όλες τις εξουσίες και όλα τα στοιχεία. Εγώ θα ήθελα να μα πει ε, καλύτερα ο κύριος Ράιτ ποια είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να την χάνουν επεξεργασία από τα κρατη και επομένως θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από την Ευρωπόλ. Πώς θα μπορέσει να υπάρξει λοιπόν η καλύτερη κατανομή των αρμοδιοτήτων στα θέματα της ε, επεξεργασίας των στοιχείων και συμφωνώ και εγώ με τον κύριο Δία στη μέρα ότι θέλουμε έλεγχο και όχι μια απλή εποπτεία σε σχέση με την Ευρωπόλ. Κυρία Ζίμπελ θέλει να πει κάτι παραπάνω. Θα ήθελα να πω στην κυρία Χόλμαερ δεν χρειάζεται να έχουμε πάντα ένα πνεύμα καχυποψίας, αλλά δεν μπορούμε όλα να τα βλέπουμε μονάχα με θετικό πνεύμα. Και εγώ πιστεύω ότι ο έλεγχος που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι επαρκής. Δεν νομίζω ότι μπορούν να θέτουμε προϋποθέσεις και να μην ελέγχουμε ή να ελέγχουμε μόνο εκ των υστέρων πώς εφαρμόζονται. Εμείς θα θέλουμε να ξέρουμε ποιες είναι οι συνθήκες, ποιες είναι οι προθέσεις και τότε να θεσπίσουμε τους κανόνες για το πώς θα λειτουργήσει η Ευρωπόλ. Εμείς πάντα θέλουμε να έχουμε την απαραίτητη εμπιστοσύνη στις αρχές ότι προφανώς θα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες μονάχα προς τον σκοπό της αντιμετώπισης του εγκλήματος και της πρόληψης. Αλλά όπως λέμε στα γερμανικά σε μια παροιμία, καλή είναι η εμπιστοσύνη, καλύτερος ο έλεγχος όμως. Όλες οι πληροφορίες λοιπόν που θα την χάνουν ανταλλαγή ή παράδοση σε τρίτους. Για μας είναι πολύ ενδιαφέρον να ξέρουμε ποια είναι αυτά τα στοιχεία, ποια στοιχεία θεωρούνται διαβαθμισμένα ή ευαίσθητα, πώς υπάρχουν οι προδιαγραφές ασφαλείας στην επεξεργασία των στοιχείων και πώς γίνεται η χρήση των νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση του εγκλήματος. Πρέπει φυσικά να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνουν οι νέες τεχνολογίες, αλλά πολλές φορές βλέπουμε ότι υπάρχει ανεπαρκής κατάρτιση του προσωπικού ή δεν, λειτουργεί, δεν λειτουργούν καλά οι διάβλοι επικοινωνίες. Ίσως λοιπόν πρέπει να ζητήσουμε πρώτα τα κρατη να κάνουν σωστά τα καθήκοντά τους στον τομέα αυτό και όχι να δημιουργούμε νέους φορείς. Αυτό δεν είναι θέμα καχυποψίας, απλώς σημαίνει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανάγκη να υπάρξει μια μεγαλύτερη σαφήνεια για να ξέρουμε ότι όλα αυτά τα οποία έχουμε αποφασίσει είναι αυτά τα οποία θα γίνουν και να μην καταλήξουμε τελικά σε μια κατάσταση πλημμυρίδας πληροφοριών τα οποία δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε και δεν ξέρουμε με ποιον ανταλλάσσονται και με ποιον όχι. Ευχαριστώ. Κυρία Χόλμαερ, θέλετε να απαντήσετε. Δεν θέλω τώρα να ξεκινήσουμε ένα διμερή διάλογο, αλλά για το θέμα της ε, καχυποψίας, εγώ είχα αγαπητή κυρία Σίμπελ να, την ευκαιρία να δω πολλά από αυτά τα θέματα και να μπω σε λεπτομέρειες και αυτό ουσιαστικά μείωσε και το επίπεδο καχυποψίας μου. Βάσει των στοιχείων λοιπόν που είχα δει εγώ δεν βλέπω ότι η Ευρωπόλ έχει καμία πρόθεση να αφαιρέσει αρμοδιότητες από τα κράτη-μέλη και να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία και τις εξουσίες στην, ε, στα χέρια της. Απλώς είναι φανερό ότι χρειάζεται και περισσότερη προσπάθεια κατάρτισης ώστε να αντιμετωπίσει τους διάφορους τομείς όπου δραστηριοποιείται. Να το πω πιο συγκεκριμένα, το κέντρο αυτό το κατά του κυβερνοεγκλήματος δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι θα αντικαταστήσει τα εθνικά κέντρα. Αντίθετα, το Ευρωπαϊκό Αυτοκέντρο χρειάζεται την αρρωγή των εθνικών κέντρων, γιατί χωρί αυτά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Εντάξει, φτάνουν όλα αυτά, λέει ο πρόεδρος. Επανερχόμεθα τώρα στους δύο φιλοξενουμένους μας. Ακούσαμε τις παρουσιάσεις τους, ακούσαμε και τα μέλη ίσως θέλουν να συμπληρώσουν κάποια πράγματα. Κύριε Γουένραϊτ, ακούσατε τις απόψεις των κρατών μελών, τα σχόλιά τους περισσότερο και όχι τόσο ερωτήσεις. Μπορεί να θέλετε να τα σχολιάσετε κι εσείς με τη σειρά. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για όλα τα χρήσιμα σχόλια. Η κυρία Ζήπελ έχει δίκιο. Είμαστε στην αρχή μια σημαντικής διαδικασίας συζήτησης και εδώ σε αυτό το βήμα αλλά και αλλού. Αυτό θα ξεκινήσει όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάσει την πρόστασή της στο τέλος του χρόνου. Αλλά ήδη σήμερα έχουμε θέσει κάποια από τα πιο σημαντικά θέματα για τον κύριο Διαστεμέρα έχει και ο ίδιος τη δική του εμπειρία, τη δική του σταδιοδρομία, ξέρει τι σημαίνει καταπολέμηση εγκλήματος και τι είναι σημαντικό. Αυτό που είναι σημαντικό λοιπόν είναι να έχουν την δυνατότητα οι ανακριτές να χρησιμοποιούν τις σωστές πληροφορίες στο σωστό χρόνο σε ένα ευέλικτο περιβάλλον όπως στα πλαίσια της χρήσης του κινητού γραφείου. Αυτό το οποίο στο οποίο αναφερόμαστε είναι μία μορφή εσωτερικής αναδιοργάνωσης και ένα streamlining της γραμματείας έτσι η Europol να γίνει πιο αποτελεσματική και να μπορούμε εμείς τα στοιχεία να τα εξετάζουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο και να προσπαθούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις παράνομες δραστηριότητες. Έρχομαι εδώ σε αυτά τα οποία είπε η κυρία Ζίπλ, ότι το Κοινοβούλιο είναι υπέρ όσο λιγότερο συστημάτων γίνεται. Και εμείς θέλουμε να ισχύει αυτό και εμείς θέλουμε να λειτουργούμε σε ένα αποτελεσματικό περιβάλλον, ιδιαίτερα σε επίπεδο αναλυτικό για τις ανταλλαγές απόψεων ανάμεσα στους δύο τελευταίους ομιλητές ή καλύτερα στις δύο τελευταίες ομιλήτριες. Αυτό το οποίο δεν αλλάζει είναι ο βασικός χαρακτήρας της δουλειάς της Europol. Εμείς εδώ στηρίζουμε αν θέλετε και βοηθάμε τα κράτη-μέλη. Δεν αναλαμβάνουμε εκτελεστικές δράσεις μόνοι μας, δεν κάνουμε εμείς προτάσεις ακόμα και στα πλαίσια του νέου κέντρου για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος. συντονιζόμαστε με τις εθνικές αρχές στο βαθμό που υπάρχει ανάγκη για μια κεντρική ευρωπαϊκή αρχή η οποία να συγκεντρώνει τις εμπειρίες, να είναι το κέντρο συλλογής πληροφοριών και εμπειριών πριν από την ανταλλαγή τους ανάμεσα στα εθνικά αντίστοιχα επίπεδα. Νομίζω ότι αλλιώς δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα σε εθνικό επίπεδο κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Αυτό θα πρέπει να διαφαίνεται και στις δυνατότητες που έχουμε να χειριζόμεθα τα μέσα, τα δεδομένα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, να προσπαθούμε να συνδυάσουμε δηλαδή ε, τα στοιχεία που προέρχονται από διάφορες χώρες που χρησιμοποιούν το ίντερνετ για να βλάψουν τις κοινωνίες μας. Για να τους παρακολουθούμε σωστά πρέπει να συλλέγουμε πληροφορίες και από τις εθνικές αρχές και γι' αυτό απαιτείται ε, πιο αποτελεσματικός μηχανισμός συλλογής των πληροφοριών. Αφού συλλέξουμε τις πληροφορίες χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για να εντοπίσουμε την εγκληματικότητα και να μπορέσουμε και εμείς με τη σειρά μας να στηρίξουμε τις προσπάθειες που κάνουν τα εθνικά, οι εθνικές υπηρεσίες. Να στηρίξουμε με τη γνώση της μίας υπηρεσίας αυτό που μία άλλη, σε μία άλλη χώρα κάνει και να καταστήσουμε ακόμα περισσότερες δυνατές παρεμβάσεις αστυνομικές από τη μία χώρα στην άλλη. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε τα μέσα για τη συλλογή των δεδομένων, για την σόρευση, αποθήκευση των δεδομένων. Αυτό γίνεται από πάρα πολλούς παροχής δεδομένων Φυσικά αυτές θα είναι κατασταλτικές η ε, ε, αστυνομικές αρχές, αλλά ιδιαίτερα στο κυβέρνο έγκλημα βλέπουμε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις ε, ιδιωτικής φύσεως οι οποίες κατέχουν πάρα πολλά ιδιωτικά δεδομένα όπως η παροχή στο διαδίκτυο κτλ. Οι εθνικές αρχές εξαρτώνται κατά πολύ από τη στενή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και θα πρέπει και εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κάνουμε το ίδιο. Τώρα σχετικά κυρία Ζήπελ με τα ευαίσθητα δεδομένα, προφανώς και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί εδώ σε επίπεδο νομικό τα ευαίσθητα δεδομένα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν πληροφορίες σαν παράδειγμα με την σεξουαλική δραστηριότητα ενός συγκεκριμένου πολίτη. Αυτό είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Εμείς ας πούμε προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την παιδοφιλία ε, στο διαδίκτυο. Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα τα οποία λαμβάνονται υπόψη σχετικά με τη σόρευση των προσωπικών δεδομένων γιατί ξέρουμε ότι είναι πολύ λίγα τα περιθώρια τα οποία έχουμε για να, να κινηθούμε νόμιμα. Όλα αυτά συμβαίνουν όμως μέσα σε αυτό το οποίο έχουμε δηλαδή ένα δίκτυο ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων αρκετά αυστηρό και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ό,τι περισσότερες δυνατότητες έχουμε για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα της συλλογή των δεδομένων. Έχουμε λοιπόν μια ε, πρόσβαση ε, θα έλεγα προνομιούχας στις βάσεις των προσωπικών δεδομένων και θα πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε με τη μέγιστη δυνατή προσοχή και επιμέλεια. Σχετικά ε, με αυτό που είπε ο κύριος Βίντενχάουζερ, τις οικονομικές μας ανάγκες. Φυσικά εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι το νέο, όπως είπε και ο κύριος ε, Διέσντε Μέρα εφόσον χρειαζόμαστε νέες, ε, νέους πόρους για να πετύχουμε τους νέους αυτούς στόχους. Στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης μπορέσαμε από το εσωτερικό της Ευρωπολ να συλλέξουμε ορισμένους πόρους προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά σε μια κλίμακα όχι επαρκή και θα πρέπει να βρούμε περισσότερους πόρους. Περιμένουμε από τις απόψεις των δημοσιονομικών αρχών ε, για τα θέματα αυτά στα πλαίσια του προϋπολογισμού του επομένου έτους. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και την Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί δείχνουν τη μέγιστη δυνατή κατανόηση για τις ανάγκες μας. Τώρα, σχετικά με την αυξημένη ροή πληροφοριών για το οργανωμένο έγκλημα και εδώ ε, για, τα, για το κόστος έχουμε κάποιες μικρές δυνατότητες αύξησης των μέσων μας. Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί και από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και από το να αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η εποχή δεν είναι πολύ εύκολη για οποιαδήποτε μορφή αύξησης του προϋπολογισμού. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ και τους ομιλητές για τις θετικές τους παρατηρήσεις και τα καλά τους λόγια. Ευχαριστώ κύριε Wainwright. Ως ε, συνήθως απαντήσατε σε όλες τις ε, παρεμβάσεις. Τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Πρίβε. Είμαι σίγουρος ότι και εσείς θα θέλετε να σχολιάσετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κάποια στιγμή μπήκα στον πειρασμό να μιλήσω γερμανικά, τελικά όμως θα επιμείνω. Θα μιλήσω αγγλικά. Ελπίζω, θα υπόσχομαι ότι θα είμαι πιο ακριβής στην ορολογία. Κατά την κατάρτιση ενός ε, νέου κανονισμού, ουσιαστικά τώρα έχουμε μια προκατακτική συζήτηση πριν από την ε, πρόταση όπως σε κάθε μέσο λοιπόν σε αυτό τον τομέα της καταπολέμησης ε, του εγκλήματος και ε, για την ασφάλεια, το, το βασικό θέμα είναι η αποτελεσματικότητα και οι εγγυήσει. Βεβαίω και θα λάβουμε υπόψη οποιαδήποτε αρχή προστασίας δεδομένων εφόσον ε, το έργο της Ευρωπόλ αφορά σε μεγάλο βαθμό την ανταλλαγή δεδομένων. Έγινε πρόταση στις αρχές ε, του έτους για την προστασία δεδομένων που δεν ε, έχει ως στόχο να αφορά άμεσα ε, τους, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά δεν θα γίνει μια νέα πρόταση από την Επιτροπή για τη νέα νομική βάση της Ευρωπόλ. Δεν θα αλλάξει τίποτα λοιπόν στις αρχές ε, για την προστασία δεδομένων. Βεβαίως ε, αυτές οι αρχές αφορούν κυρίως τον ιδιωτικό τομέα. Αλλά ξέρουμε ακριβώς ε, τι πρέπει να κάνουμε για την νέα πρόταση νομικής βάσης για την Ευρωπόλη. Πρέπει να ορίσουμε τα κατάλληλα εχέγγυα. Έως τώρα πάντως έχουμε δει ότι η Ευρωπόλ έχει πολύ ψηλά πρότυπα. Εξάλλου, το να λέμε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει με μεγαλύτερη προσοχή και επιμέλεια να δίνουν ε, δεδομένα προς την Ευρωπόλ, αυτό για μένα είναι ένα σημείο που αφορά την αποτελεσματικότητα, όχι την προστασία δεδομένων. Οι κανόνες πρέπει να είναι ίδιοι, ανεξάρτητα από τον όγκο ε, των πληροφοριών που ανταλλάσσονται. Ένα άλλο θέμα που θα συζητηθεί σίγουρα είναι το πώς ε, η Ευρωπόλ θα μπορούσε να ανταλλάζει πληροφορίες με τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό βέβαια πρέπει να γίνει πάντα ε, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και, και την ασφάλεια, όχι βεβαίως με γνώμονα το συμφέρον των ε, ιδιωτικών επιχειρήσεων. και ακούσαμε πολλές διαφορετικές απόψεις και ακούμε ε, για το κατά πόσο αυτή η ε, εποπτική δομή θα πρέπει να συνεχιστεί ή αν θα πρέπει ε, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων να αναλάβει την Ευρωπόλ. Σε αυτό το θέμα υπάρχουν ριζικές διαφωνίες. Και πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη στην πρότασή μα. Για το EC3, αυτό το κέντρο που αναφέραμε προηγουμένως, σας ε, συνιστώ να διαβάσετε την ανακοίνωση ε, της Επιτροπής του Μαρτίου. Ε, έτσι μπορούν να λυθούν κάποιες απορίες και προβληματισμοί που αναφέρθηκαν εδώ σήμερα. Δεν υπάρχει πρόθεση να συγκεντρωθεί, να μονοποληθεί το έργο της Ευρωπόλ. Αυτό περιγράφεται πολύ καλά στην ανακοίνωση. Δεν είναι πρόταση νομικής πράξη, γιατί όπως είπε και ο Ρόμπ, αυτό είναι θέμα εσωτερικής αναδιάρθρωσης. Και βεβαίως πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να βρούμε τους απαραίτητους πόρους με εξοικονόμηση πόρων ε, μέσα από τον ε, οργανισμό αλλά και μέσω επιπρόσθετων πόρων. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις? Αν όχι, θα σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τον Διευθυντή της Ευρωπόλ, Ρόμπ Wainwright. Θα σας ξαναδούμε βεβαίως. Ευχαριστούμε και τον κύριο Πρίμπε που βεβαίως ε, μας έρχεται συχνά και συμμετέχει στις ε, συναντήσεις μας. Το τελευταίο θέμα της ε, πρωινή συνεδρίασης ε, έχει προγραμματιστεί για τις 12. Η κυρία Ντάνα και η συγγήτρια δεν είναι εδώ, επομένως προτείνω να κάνουμε διάλειμμα 25 λεπτών. we go. Φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο, σημείο 25, πολιετές πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Η συγγήτρια είναι η συνάδελφος κυρία Ντανόκα. Έχουμε το πολιετές πλαίσιο λοιπόν με τους τομείς στους οποίους η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία θα προχωρήσει στη συλλογή δεδομένων για τα επόμενα πέντε χρόνια από το 13 μέχρι το 17. Όπως γνωρίζετε, το υπάρχον πλαίσιο λύγει στο τέλος του χρόνου και υπάρχει δυνατότητα για το Συμβούλιο και την οποία τρόποι εφόσον το επιθυμούν να πάρουν το λόγο. βασική ιδέα αυτής της ανταλλαγής απόψεων είναι και να τεθεί μια προθεσμία χρονική για την κατάθεση των τροπολογιών η οποία προβλέπεται για την 25η Σεπτεμβρίου κανονικά. Κυρία Στανόκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχετε καλύψει ένα μέρος του έργου μου με την παρουσίαση των στοιχείων του θέματος αυτού. Είναι γεγονός ότι το πενταετές πολυετές πλαίσιο εκπνέει το 2017 και πρέπει να εκπονηθεί το νέο πολυετές πρόγραμμα. Υπήρξαν πολλές προτάσεις λοιπόν γι' αυτό στην αιτιολογική έκθεση μπορείτε να βρείτε την σύγκριση του προηγούμενου πολιετούς προγράμματος το οποίο είναι ακόμα ενισχύει αλλά θα εκπνεύσει στο τέλος του χρόνου την πρόταση της, της του φορέα αυτού για τα θεμελιώδη δικαιώματα για το επόμενο πενταετές πρόγραμμα και περιλαμβάνει ορισμένα σημεία όπως είναι η συνεργασία των δικαστικών αρχών, η συνεργασία των αστυνομικών, η αντιμετώπιση των διακρίσεων, όπως λέει το άρθρο 21 της Χάρτας Θεμελιώδων Δικαιωμάτων. Έχουμε επίσης την πρόταση της Κομισιόν και η Κομισιόν προτείνει μεταξύ άλλων και αναφέρεται εκπεφασμένα στο θέμα των διακρίσεων προτείνει την αστυνομική και δικαστική συνεργασία και άλλα θέματα. Δυστυχώς προτάσεις αυτές δεν έγιναν απόλυτα δεκτές από το Συμβούλιο. Κατά την ε, εκπόνηση της εκθεσής μας Συναντήσαμε τους εκπροσώπους του Συμβουλίου, της Δανικής Προεδρίας συγκεκριμένα. Μας ε, ζήτησαν συγγνώμη, αλλά είπανε δεν έχουμε συνένεση στο Συμβούλιο για ένα αριθμό προτάσεων. Ιδίως ό,τι αφορά την αστυνομική και δικαστική συνεργασία. Μπορείτε να δείτε ότι οι θεματικοί τομείς που προτείνονται από το Συμβουλίο είναι πιο συντετμημένοι και σύντομοι από αυτούς που πρότεινε το Διοικητικό Συμβούλιο και η Κομισιόν και δεν συμπεριλαμβάνουν την δικαστική και την αστυνομική συνεργασία. Ούτως εχόντων των πραγμάτων, ποια μπορεί να είναι η θέση μας, η θέση του Κοινοβουλίου. Βέβαια σε άλλες συνθήκες εγώ θα προσκαλούσα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην συνενέσει και να αναζητήσει μια καλύτερη λύση για το 54 αυτό πρόγραμμα. Βρισκόμαστε όμως σε μια κατάσταση που χρειάζεται νέες θεματικές περιοχές εργασίες ο φορέας αυτός αν δεν υπάρχει ένα νέο πολίτες ε, πρόγραμμα ενισχύει από την αρχή του 2013 ο φορέας αυτός δεν θα μπορεί να πράξει τίποτα παρά μόνο αν υπάρχει μια ειδική αίτηση από κάποιο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι αυτό το οποίο θα θέλαμε βέβαια. Και ως εκ τούτου εκφράζω στην αιτιολογική μου έκθεση πολλά σημεία που δείχνουν την δυσαρέσκειά μας, την έλλειψη ικανοποίησης από την πλευρά του Κοινοβουλίου και ελπίζω θα τα υποστηρίξει η Επιτροπή μας. Εκφράζω τη λύπη μας για το γεγονός ότι δεν υπήρξε συμφωνία στο Συμβούλιο σε σχέση με τις νέες θεματικούς τομείς της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας και της αναγνώρισης ε, της αμοιβαίας σε ποινικά θέματα. Επίσης εκφράσαμε και την ανησυχία μας για το μήνυμα που δίνει το Συμβούλιο με την έλλειψη απόφασης που δεν ενισχύει την ε, πρόθεση των θεμάτων αυτών που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα λοιπόν του πολιετούς πλαισίου αυτού στο, στο σχέδιο αυτό προτείνεται να εξαιρεθούν από τα θέματα διακρίσεων περιπτώσεις που εμπλέκουν μια εθνοτική μειονότητα. Το βρίσκουμε αυτό απαράδεκτο. Λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αρχές του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αξιών και αυτό συμπεριλαμβάνει τα άτομα τα οποία ανήκουν σε μειονότητες, είναι το άρθρο 2 λαμβανωμένων υπόψη όλων αυτών, η έκθεση αναφέρει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει την έκθεσή του στο νέο πολιετές πλαίσιο, αλλά εκφράσουμε την ελπίδα μας ενδιαμέσως ότι η Κομισιόν θα επανεξετάσει τους στόχους που θα πρέπει να εξυπηρετήσει αυτός ο φορέας και ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο θα είναι έτοιμο να προχωρήσει σε μια συμφωνία μέσα σε αυτό το πλαίσιο για την συμπερίληψη της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας σε ποινικά θέματα τουλάχιστον σε αυτούς τους θεματικούς τομείς. Και ελπίζουμε το Συμβουλίο θα προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτά για την αιτιολογική έκθεση και θα ήθελα εν κατακλείδη να ευχαριστήσω τους σκιοδησίτες για τις συναντήσεις μαζί μου και συναντήσεις με το Συμβούλιο, παρουσία και της Κομισιόν. Να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Κομισιόν και τους συνεργάτες μου, τον Αλεξάνδρου Βίτροφ και τον Τζόσα Κάντας, που με βοήθησαν να συντάξω αυτήν την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην Επιτροπή ή στο Συμβούλιο. Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά την κυρία Στάνοκα. Ε, για το έργο της και για το, το σχέδιο συστάσεων που προτείνει το Κοινοβούλιο να ε, εγκρίνει το σχέδιο απόφασης ε, που, που έχει παρουσιαστεί από το Συμβούλιο. Όπως γνωρίζετε, είχαμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με την κυρία Συγητρία. Η Επιτροπή έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να ε, λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ε, για την συμπερίληψη των θεματικών τομέων ε, της αστυνομική και δικαστικής συνεργασίας ζητήματα ποινικού δικαίου. Για την Επιτροπή μετά την συνθήκη τη Λισαβόνα, έπρεπε να συναχθούν κάποια συμπεράσματα. Πλέον δεν υπάρχουν πυλώνες Κάποιος ε, οργανισμός λοιπόν πρέπει να είναι σε θέση να ε, εργαστεί σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από το ενωσιακό δίκαιο. Όμως ε, βλέπουμε ότι παρόλες τις προσπάθειες δεν κατέστη δυνατό στο Συμβούλιο να ε, επιτευχθεί η ομοφωνία. Όπως ξέρετε αυτό το σχέδιο απόφασης για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο βασίζεται στο άρθρο 372 της συνθήκης και απαιτείται ομοφωνή απόφαση. Διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν δυνατό αυτό. Ε, με λύπη μου το λέω και χρειάζεται και πάλι ένα ε, συμβούλιο και διαπιστώνεται, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν καλύπτεται αυτός ο θεματικός τομέας από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ωστόσο, όπως είπε η κυρία Στανόκα, είναι σαφές ότι είναι απαραίτητο για τον οργανισμό να έχει ένα Πολιετέ πλαίσιο που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013. Θα ήταν ε, πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον οργανισμό αν δεν υπήρχε τέτοιο ε, πολιετές πλαίσιο, γιατί τότε ο οργανισμός δεν θα μπορούσε να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο εργασιών του, ε, το οποίο το υιοθετεί εντελώς ανεξάρτητα, όπω γνωρίζετε, και το υλοποιεί σε ένα πολιετές πλαίσιο. Εάν δεν υπάρχει πολιετές πλαίσιο, τότε ο οργανισμός δεν μπορεί να υλοποιήσει το πρόγραμμα εργασιών του. Μεγάλο λοιπόν το πρόβλημα και συμφωνούμε απόλυτα με την εισηγήτρια Παρόλο που λυπούμεθα που ε, δεν υπάρχουν αυτοί οι θεματικοί τομείς στο σχέδιο απόφασης, θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, τεθεί σε ισχύ αυτό το ε, πλαίσιο, το πολιτές πλαίσιο, την 1η Ιανουαρίου 2013. Ευχαριστούμε λοιπόν την εισηγήτρια που πρότεινε στο Κοινοβούλιο να υιοθετήσει την απόφαση του Συμβουλίου, ακόμα και αν ε, δεν ήταν η ευκταία ούτε από την Επιτροπή ούτε από την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την Επιτροπή. Να δώσουμε το λόγο τώρα στα μέλη. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Γκάλ. Thank you, Chair. I was the... Ευχαριστώ. Ήμουν σκιώδη συγγήτρια για αυτή την έκθεση εκ μέρους του ΕΛΚ. Ε, συμφωνώ πολύ με την συγγήτρια Αυτή η απόφαση πρέπει να ε, ληφθεί μέσω διαδικασιών του, του Συμβουλίου. Επομένω, ε, το Κοινοβούλιο μπορεί να απαντήσει θετικά ή αρνητικά. Το πολιετέ πλαίσιο για τον οργανισμό αυτό 2013-2017 θα έρθει του χρόνου. Ο οργανισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς τη θετική μας γνώμη. Επομένως, συμφωνώ ότι πρέπει και εμείς ε, ε, να υιοθετήσουμε αυτό το νέο πλαίσιο μέχρι τα τέλη του 2012. Επίσης, και εγώ λυπούμε που ε, το Συμβούλιο δεν προσέθεσε την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ζητήματα ποινικού δικαίου. Θεωρώ και εγώ ότι αυτό πρέπει να αλλάξει στο μέλλον. Αυτά. Thank you. Ευχαριστούμε. Κυρία Ζέροκα. Thank you very much. Ευχαριστώ, Να συμφωνήσω με την άποψη της κυρίας Ντάνουκα. Γιατί πράγματι η υπηρεσία αυτή παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε πάρα πολλούς τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε ένα κεκτημένο λοιπόν, αλλά πιστεύουμε ότι τα τελευταία χρόνια ή μάλλον τα επόμενα πέντε χρόνια το να συνεχιστεί ακριβώς αυτό που προηγήθηκε δεν επαρκεί και αν κοιτάξει κανείς κάποια επιμέρους θέματα θα δει ότι πράγματι ξεκίνησαν πολύ καλά κάποια θέματα όπως η στρατηγική των Ευρωπαϊκών Τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Αλλά όταν βλέπει κανείς κάποια συγκεκριμένα επιμέρους θέματα, βλέπουμε ότι οι δυνατότητες της υπηρεσίας είναι μικρότερες από αυτές τις οποίες επιθυμούσαμε. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει με ποιο τρόπο οι χώρες σέβονται τις ε, ρυθμίσεις οι οποίες έχουν συμφωνηθεί. Συμφωνώ επίσης με αυτά τα οποία λέτε ότι η ενσωμάτωση σαν παράδειγμα των Ρωμαίων αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επαναξεταστεί πλήρως. Υπάρχουν και άλλοι τομείς τους οποίους θα πρέπει να προσπαθήσει η υπηρεσία να καλύψει και ελπίζω συνεργαζόμενοι στενά με την υπηρεσία μπορούμε πράγματι με τις κατάλληλες επαγγελματικέ συμφωνίες να καλύψουμε τις ανάγκες. Συμφωνούμε λοιπόν με την εισηγήτρια περιμένοντας όπως είπα πάντα και κάποιες περαιτέρω εξελίξεις. Ευχαριστώ κύριε Γιαρόκ. Η κυρία Βεργιά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς δεν έχω παρακολουθήσει το σύνολο της ε, συνάντησης που είχαν διοργανώσει τρεις συγητές. Εγώ συμμεριζόμαι απόλυτα την ε, πρόοδο που έχει επιτευχθεί μάλλον τα σχόλια σε σχέση με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στους κόλπους του Συμβουλίου, ιδίω όταν ξέρουμε ότι στον τομέα αυτό είναι σημαντικέ παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η έκθεση που έχουμε εγκρίνει την προηγούμενη εβδομάδα για την υπόθεση και για μα καταδεικνύει την αλήθεια αυτών των λεγόμενων. Μόνο ένα ερώτημα έχω να θέσω στην εισηγήτριά μα, επειδή στην έκθεσή της λέει ότι ελπίζει ότι πριν από την οριστική έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσαν να υπάρξουν εξελίξεις στους κόλπους του Συμβουλίου. Τι εννοεί ακριβώς. Εάν εγκρίνουμε την έκθεση της όπως έχει τώρα, μήπως χάνουμε τη δυνατότητα άσκησης πίεσης προς το Συμβούλιο και προς την Κομισιόν. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θέλω να θέσω. Κατά τα άλλα συμμεριζόμαι απόλυτα την κατεύθυνσή της. Σας ευχαριστούμε κυρία Βερζιά. Ελήψη άλλων σχολείων. Θα ξαναδώσω το λόγο στην εισηγήτρια, στην κυρία Στάνοκα. Μάλιστα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και όλους φυσικά τους συναδελφούς που έλαβαν το λόγο και υποστηρίξη την προσέγγιση μου. Κυρία Βεζιά, συμφώνω μαζί σας. Εάν εμείς δεν δίναμε την έκκλησή μας και απορρίπταμε το νέο πρόγραμμα θα ήταν μια μορφή άσκησης πίεσης προς το Συμβούλιο. Δυστυχώς όμως Όταν είναι κανείς στην πολιτική, είναι πάντα μεταξύ σφύρας και άκμονος. Πρέπει να κάνει κανείς μια επιλογή μεταξύ μεταξύ προβληματικών καταστάσεων και πρέπει να αποδηθεί και σε θυσίες. Και είχαμε και πολλές διαβουλεύσεις με το Φορέα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και θεωρούν ότι η δεύτερη επιλογή, το να μην δώσουμε δηλαδή την έγκριση μας στο νέο πρόγραμμα, θα οδηγούσε σε πλήρη μπλοκάρισμα του έργου του Φορέα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, η πρότασή μας εξακολουθεί να συνεχίσουμε το διαλόγο και η κυρία Γκάλ που ήταν συγγήτρια για τον φορέα αυτό όταν ξεκίνησε το 2007 θεωρούμε ότι πρέπει να συζητήσουμε τον νέο κανονισμό επί τη βάση μιας νέας νομικής βάσης και μετά μπορούμε να επαλέθουμε και κυρία Γερόκα σας ευχαριστώ επειδή αναφέρατε την ε, λύπη σας για την ε, όχι ικανοποιητική διατύπωση στο θέμα της ενσωμάτωσης των Ρωμά. Μεταξύ των θεματικών τομέων θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη διατύπωση στο θέμα αυτό. Και υπήρχε στο παρελθόν ένα πρόγραμμα εργασίας και για τα θέματα αυτά και η συνεργασία μας με το Συμβούλιο δεν ευνοήθηκε από την αλλαγή Προεδρίας τον Ιούλιο. Η Κυπριακή Προεδρία δεν είχε συμμετάσχει πλήρως στις συζητήσεις και μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει κίνηση στο Συμβούλιο. Και επομένως η πρότασή μου είναι να κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις κριτικού χαρακτήρα σε σχέση με τη συμπεριφορά του Συμβουλίου και ελπίζω θα καταθέσετε και τροπολογίες αν δεν είστε ικανοποιημένοι με το επίπεδο επικρίσεων που θα ενσωματώσω στην έκθεσή μου. Θέλω να ευχαριστήσω και τη γραμματεία της Επιτροπής ε, Λίμπε, η Μαρία και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε αυτή τη γνωμοδότηση και να την διαβιβάσουμε και στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Κυρία Βερζιά, θέλετε το λόγο. Αλλά, ναι, ναι, κύριε Πρόεδρε. Απλώς ίσως δεν έγινα κατανοητή από την κυρία Ζτανόκα. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά που λέει στην παραγραφή της, είναι περισσότερο θέμα στρατηγικής και χρονικής αλληλουχίας. Δεν ζητάω την απόρριψη του προγράμματος. Λέω απλώς μήπως αναστείλουμε τη διαδικασία ψηφοφορίας της έκθεσης αυτής για να ασκήσουμε πίεση, μήπως έλθουν και κάποιες προτάσεις. Καταλαβαίνω το πρόβλημα, δεν ζητώ να απορριφθεί αυτή η πρόταση και να κάνουμε αδύνατο το έργο αυτού του φορέα που είναι πάντα χρήσιμο ανεξάρτητα από τα όρια που του θέτει το Συμβουλίο. Το κατανοήσαμε. Ναι, δυστυχώ λέει κυρία Στανόκα. Σε τρεις ε, μήνες τελειώνει το έτος και το χρονοδιάγραμμά μας έχει υπολογιστεί ώστε να έχουμε για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε εγκαίρως. Δεν μπορούμε όμως δυστυχώς να, να βάλουμε περαιτέρω την ψηφοφορία λόγω αυτού του χρονικού ορίου. Και μετά αλλάζει η Προεδρία. Η Ιδανική Προεδρία έκανε όλες τις απαραίτητες προσπάθειες, αλλά το αποτέλεσμα που προέκυψε είναι αυτό που γνωρίζετε. Ακόμα και με την πρόταση να αφαιρεθούν τα δικαιώματα των μειονοτήτων, και αυτό είναι σκανδαλώδες πιστεύω. Okay, we thank you again, Mrs. Στανόκα. Αυτά για σήμερα. Ερχόμαστε στο τέλος της συνεδρίασης. Τρεις η ώρα συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας. Αλλά θα ήθελα να σας πω ότι για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, για το πολιετές πλαίσιο για την, φορέα θεμελιωδών δικαιωμάτων, να έχουμε υπόψη ότι βάσει των χειμένων κανόνων για το θέμα αυτό, θα έχουμε μια διαδικασία σύμφωνης γνώμης. Μόνο διαδικαστικού χαρακτήρα τροπολογίες λοιπόν είναι παραδεκτές για την έκθεση αυτή. Και αυτό θα πρέπει να το έχετε υπόψη Δεν μπορούμε να έχουμε τροπολογίες προς το περιεχόμενο, απλώς διαδικαστικές τροπολογίες. Και αυτό αφορά και την αιτιολογική έκθεση. Τροπολογία για Τροπολο... Προθεσμοί για τροπολογίες είναι, είναι την 3η 25 Σεπτεμβρίου. Τρεις η συνεχίζουμε την εργασία μας.